εγκριθεί όπως έχει. Προχωρούμε στη συζήτηση. Προετοιμασία για τη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον λόγο στον κύριο Λετσκεβίτσιου. Uh, uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξότιμοι Ευρωβουλευτές, Πρόεδρε Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ χαίρομαι που σήμερα το πρωί συμμετέχω στη συζήτηση αυτή σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη επόμενη εβδομάδα. Υπάρχουν πολλά πράγματα στην ημερήσια διάταξη, μεγάλο εύρο θεμάτων που έχουν να κάνουν με την άμυνα, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, την Οικονομική και την Κοινωνική Πολιτική. Θα αρχίσω με την άμυνα. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει συζήτηση για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Και αυτό έρχεται σε μια πολύ καλή στιγμή. Τέσσερα χρόνια αφού το άρχισε να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας. Και λαμβάνει η χώρα επίσης σε μια στιγμή που υπάρχει και κάποια απογοήτευση όσον αφορά τις αξίες της Ευρώπης. Έτσι έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία να δείξουμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρώπης ή, για να το πω διαφορετικά, να δείξουμε ότι το κόστος του να μην έχουμε Ευρώπη είναι πολύ μεγαλύτερο. Και ξέρω ότι είναι θέματα τα οποία απασχολούν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ. Αυτό φάνηκε και από τη συζήτηση που έγινε με τα Εθνικά Κοινοβούλια το Δεκέμβριο του 2013. Ο προπολογισμό της άμυνας μειώνεται και υπάρχει κάποιος κατακαιρματισμός. Συνεπώς, αν τα κράτη-μέλη εναρμονίσουν τις ε, απαιτήσει τους όσον αφορά τις στρατιωτικές ικανότητες, τότε μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους πολύ πιο αποτελεσματικά και μπορούν να αποφασίσουν από κοινού να χρησιμοποιήσουν και να συντηρήσουν τον εξοπλισμό που διαθέτουν και έτσι να έχουν πολύ καλύτερη αποτελεσματικότητα από ό,τι θα είχαν από μόνοι τους σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν ε, τέτοια παραδείγματα όπως ο ανεφοδιασμός εν πτήση, το οποίο είναι μια Πολύ καλή απόδειξη. Καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί να έχει στη διάθεσή της τον ε, απαραίτητο εξοπλισμό και όλα τα αεροπλάνα που χρειάζονται για να γίνει αυτός ο ανεφοδιασμός σε πτήση. Έτσι λοιπόν, με στενή συνεργασία μεταξύ μας, μπορούμε να αυξήσουμε την ικανότητά μας, να μειώσουμε το κόστος και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Και αυτό είναι αλήθεια και για την αμυντική μας βιομηχανία διότι η τεχνολογική και η βιομηχανική μας βάση είναι κατακαιρματισμένη. Αν λοιπόν η Ευρώπη θέλει να διατηρήσει τη στρατηγική της αυτονομία και να διασφαλίσει τον ανεφοδιασμό, τότε χρειάζεται δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επιπλέον πρέπει να δημιουργήσουμε μια αμυντική βιομηχανία πιο ανταγωνιστική και πιο ολοκληρωμένη, κάτι το οποίο θα βοηθήσει και σε δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση, καινοτομία και ανάπτυξη. Βέβαια, είναι οι επικεφαλεί κρατών και κυβερνήσεων οι οποίοι θα εξετάσουν τη συνολική εικόνα και θα αποφασίσουν για κατευθυντήριε γραμμέ. Πώ μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν συνολικό τρόπο να ανταποκριθεί στι τόσο γρήγορε εξελίξει που έχουμε την ευρωπαϊκή στρατηγική στο γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε και πώς θα αντιμετωπίσω θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, κυρίως την ενέργεια, τον κυβερνοχώρο ή τη θάλασσα. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες της και να προσφέρει ασφάλεια, ειρήνη μαζί με τους εταίρους της κλειδί. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα καθορίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτεραιότητες γύρω από τρεις άξονες. Πρώτον, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της προβολής και του αντικτύπου, το συνεπείο μπορεί να έχει η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει μαζί με έναν συλλεκτικό τρόπο πολιτικές, να τη συνδυάσει δηλαδή πολιτικές και εργαλεία, είτε πρόκειται για τη διπλωματία, την ασφάλεια, την άμυνα, τα οικονομικά, το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη δικαιοσύνη. Όλα αυτά μπορούν παρατέρω να βελτιωθούν. Έπειτα υπάρχει το θέμα των ικανοτήτων Άμυνα. Έχω ήδη αναφέρει ότι η συνεργασία μεταξύ χωρών μελών είναι ζωτική σημασία, διότι έτσι μπορεί να έχουμε πιο συντονισμένη δράση, σχεδιασμό αμυντικό, ικανότητε ανάπτυξη και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Τέλο, έρχομαι στην ενίσχυση τη αμυντική μα βιομηχανία. Πρέπει να βελτιώσουμε τι συνέργειε που υπάρχουν ανάμεσα στο στρατιωτικό τομέα και τον μη στρατιωτικό τομέα στην έρευνα. Μπορούμε να μειώσουμε το κόστος, να αναρμονίσουμε τη ζήτηση και να ενισχύσουμε τη διαλειτουργικότητα αναπτύσσοντας αμυντικές βιομηχανικές προδιαγραφές και διαδικασίες αδειοδότησης, χωρίς να γίνονται επικαλύψεις. Αυτό θα μας βοηθήσει να δώσουμε καλύτερη πρόσβαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν βέβαια στοιχείο κλειδί για την ανάπτυξη των αγορών αυτών. Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, διαπιστώνουμε μια σταδιακή ανάκαμψη στην οικονομία μα. Σιγά σιγά επιστρέφει η ανάπτυξη. Όμω τα ποσοστά ανεργία είναι ακόμα πολύ ψηλά, οπότε δεν μπορούμε να εφησυχαστούμε. Χρειάζονται περισσότερε προσπάθειε. Γι' αυτό είναι ζωτική σημασία οι ηγέτε κρατών και κυβερνήσεων να κάνουν ό,τι μπορούν για να ενισχύσουν ε, πολιτικέ ενίσχυση τη απασχόληση. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξετάσει και το θέμα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Θα υπάρξει μια αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης στις χώρες μέλη και στην Ευρωζώνη βάσει της ε, ετήσιας έκθεσης για την ανάπτυξη του 2014 που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Νοεμβρίου. Θα συνεχιστεί επίσης και η δουλειά για την ενίσχυση του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής. Επιτρέψτε μου να σας πω δύο λόγια για αυτό το τελευταίο. Όπως γνωρίζετε ήδη τα τελευταία τρία χρόνια, το πλαίσιο για την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύθηκε με στήριξη ιδιαίτερη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που μόλις ξεκίνησε για το 2014 συγκεντρώνει τις διάφορες τάσεις οικονομικής διακυβέρνησης μέσα σε μια πιο συνεκτική διαδικασία. Πρέπει όμως να υπάρξει ενίσχυση της αποτελεσματικότητας παρετέρω και του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των χωρών μελών στην Ευρωζώνη. Και αυτό θα γίνει εφόσον οι χώρες μέλη ενστερνιστούν ακόμα περισσότερο και εφαρμόσουν τις συστάσεις σχετικά με την μεταρρύθμιση που οδηγεί στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Γι' αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου θα επικεντρωθεί σε θέματα συμβατικών ρυθμίσεων και μηχανισμών αλληλεγγύης. Οι συμβατικές ρυθμίσεις και οι σχετικοί μηχανισμοί αλληλεγγύης θα διευκολύνουν και θα στηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την αίσθηση του ότι είναι κτήμα μας όλα αυτά, την αποτελεσματικότητα, την ε, νομιμότητα και την λογοδοσία. Θα προχωρήσουμε με συγκεκριμένες διαδικασίες την επόμενη εβδομάδα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο περιμένουμε να αποφασίσει για τις αρχές που θα διευκολύνουν τις ρυθμίσεις αυτές. Βέβαια, η οικονομική μεταρρύθμιση είναι προς το συμφέρον των χωρών μελών. Παρ' όλα αυτά, είναι δύσκολο να αξιολογηθούν τα κέρδη άμεσα. Γι' αυτό θέλουμε οι συμβατικές αυτές ε, ρυθμίσεις να συνδυαστούν με οικονομικά κίνητρα, τα οποία ονομάζουμε μηχανισμούς αλληλεγγύης. Και αυτό και γι' αυτό θέλουμε να σχεδιάσουμε τα κατάλληλα εργαλεία για την οικονομική αυτή στήριξη. Στόχος είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποφασίσει για τα κύρια στοιχεία τόσο όσον αφορά τι συμβατικέ ρυθμίσει, όσο και του μηχανισμού αλληλεγγύη. Επιτρέψτε μου τώρα να ολοκληρώσω για αυτό το σημείο προσθέτοντας λίγα λόγια για την κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και την ολοκλήρωση της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Όσον αφορά την κοινωνική διάσταση της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να επιβεβαιώσει την απόφαση που έχει ήδη ληφθεί όσον αφορά το βαθμολόγιο για την απασχόληση και τους κοινωνικούς δείκτες. Στόχος είναι το βαθμολόγιο αυτό να χρησιμοποιηθεί στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2014. Όμως η ανάλυση των κοινωνικών δικτών δεν θα πρέπει να αποδυναμώσει τη μακροοικονομική ισορροπία. Η σχετική διαδικασία πρέπει να διατηρηθεί για να αποφευθούν ακριβώς οι μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία της ΟΝΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίση θα ασχοληθεί με την πρόοδο και την ολοκλήρωση τη Τραπεζική Ένωση. Κάτι το οποίο αποτελεί προτεραιότητα, διότι είναι πολύ σημαντικό προκειμένου να προληφθούν άλλε κρίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Με την έγκριση του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού έχει επιτελεστεί παρετέρω έργο για την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής της Τραπεζικής Ένωσης. Η Λιθουανική Προεδρία εργάζεται σκληρά προκειμένου να επιτευχθεί μια γενική προσέγγιση όσον αφορά τον ενιαίο μηχανισμό επίλυσης κρίσεων μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Χτες στο ΕΚΟΦΗΝ συζητήθηκε ακριβώς αυτό το θέμα και όπως έχω ήδη πει κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να γίνει πραγματικότητα πριν από τα τέλη της χρονιάς αυτής. Ξέρω ότι και εσείς συμφωνείτε μαζί μας για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα και θέλετε και εσείς να επιτευχθεί συμφωνία πριν από τα τέλη της θητείας αυτής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίση θα αξιολογήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο του 2012 στα πλαίσια των πράξεων 1 και 2 της ενιαίας αγοράς, όπως επίσης και στα πλαίσια τη συμφωνία για την απασχόληση των νέων και την χρηματοδότηση της οικονομίας. Είναι και αυτά θέματα τα οποία θα βοηθήσουν να επιστρέψει η ευημερία και η απασχόληση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ασχοληθεί επίση με το θέμα τη μετανάστευση στην Μεσόγειο μετά από το τραγικό ατύχημα που είχαμε στι ακτέ τη Λαμπεντούζα. Για να αποφύγουμε νέε τέτοιε καταστροφέ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο ζήτησε να υπάρξει μια task force από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα εντοπίσει δράσεις κατά προτεραιότητα για να μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ευρωπαϊκές πολιτικές και τα εργαλεία μας όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά το συντομότερο δυνατό. Και τον Ιούνιο θα συζητηθεί επίση και το θέμα του χώρου ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Την επόμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ασχοληθεί με αποφάσει προκειμένου να συνεχιστεί το έργο τη Task Force αυτή και οι και συζητήσει έγιναν επίση και από του Υπουργού Δικαιοσύνη την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, θα εξετάσουν επίσης και το θέμα της διεύρυνση την επόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπω ε, επίση, όπω γίνεται συνήθω τον Δεκέμβριο, θα έχουμε και εκθέσεις του Συμβουλίου Ενέργειας όσον αφορά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για την εσωτερική αγορά ενέργεια και τις εξελίξεις από το 2011 και μετά σχετικά με την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Αυτές οι εκθέσεις θα βοηθήσουν να συνεχιστεί το έργο μας όσον αφορά τον τομέα της έρευνας που αποτελεί στοιχείο κλειδί για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη και ασφάλεια. Πρόεδρε, το Συμβούλιο αυτό θα αποτελέσει ένα βήμα παραπάνω για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της ε, ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Ε, προσβλέπουμε σε επικοδομητικές συζητήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Επιτροπός Σεύκοτς, εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότομη μέλη. Ο Κύριε ο πρόεδρος Μπαρόζο, και θέλετε να παρήσατε εδώ γιατί τόσο σημαντική ε, συνάντηση, αποφάσισε να, πάρει, να συμμετέχει στην ε, κηδεία του Νέλσονα Μαντέλα ε, μια σημαντική πολιτική μορφή. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να σα παρουσιάσω τις, ε, την αξιολόγηση που έχει κάνει η Επιτροπή. Του προηγούμενου 12 μήνε το μήνυμα τη Επιτροπή ήταν σαφώ το παρακάτω. Σημαντικές προσπάθειες ε, ό,τι αφορά την εξυγίαση, τη σταθεροποίηση των αγορών αλλά και την ενεργή αλληλεγγύη κατεβλήθησαν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν καταφέρουμε να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες δίχως άλλο θα επιτύχουμε στην απάντηση στην κρίση καταβάλουμε προσπάθειες και αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τα αποτελέσματα. Οι οικονομικοί δείκτες δείχνουν μία μικρή ανάκαμψη. Η κατάσταση σε όλες τις χώρες έχει βελτιωθεί και έχει σταθεροποιηθεί θα, δεν θα πρέπει να, δούμε, να ξεχνάμε τι έγινε στην Ιρλανδία. Είναι δύσκολο να φανταστούμε ένα σαφέστερο μήνυμα προς τους πολίτες της Ιρλανδίας, αλλά και προς τους πολίτες όλης της Ευρώπης, αλλά και στις ε, οικονομικές χρηματοπιστωτικέ αγορές. Οι προσπάθειες ε, της Ιρλανδίας ε, αποφέρουν κακούς. Αυτός, αυτός, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποτίσουμε φόρο τιμή στους Ιρλανδούς και στην πολιτική τους ηγεσία. Το Ιρλανδικό παράδειγμα μας δείχνει ότι ότι αν υπάρξει στήριξη και ανάληψη ευθυνών, τότε θα δοθεί μια σωστή απάντηση. Αυτή είναι μια ενθάρρυνση και για άλλες χώρες που βρίσκονται ε, σε αυτά τα προγράμματα. Η Επιτροπή έχει τη βεβαιότητα ότι οι προσπάθειες, οι κοινέ προσπάθειες, δίχως άλλο θα αποφέρουν καρπούς. Η ε, Λετωνία είναι μια άλλη περίπτωση της εμπιστοσύνη στο νόμισμά μας. Το 2013 ήταν καθοριστική χρονιά σε αυτή την κρίση. Αγαπητά μέλη, το 2013 ήταν καθοριστική χρονιά και για άλλους λόγους. Καταφέραμε να υιοθετήσουμε ένα πολιετές πλαίσιο. Εγώ σκέφτομαι τις προσπάθειες που κάναμε για έναν ενιαίο μηχανισμό εποπτείας στον τραπεζικό τομέα. Έχουμε καταβάλει προσπάθειες για να ε, μεταρρυθμίσουμε την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Έχω τη βεβαιότητα ότι ο συντονισμός των εθνικών προπολογισμών γίνεται όλο και καλύτερος. Θα πρέπει όμως να διατηρήσουμε τις προσπάθειές μας. Η ανάκαμψη δεν μπορεί να αφορά μόνο λίγους. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί η ανεργία που αποτελεί πραγματικότητα για πολλές χώρες. Δεν μπορούμε ε, να αφήσουμε ημιτελές το έργο μας. Θα ήθελα να σας στείλω για μία ακόμα φορά το μήνυμα του, ε, της Επιτροπής. Ε, αξιότιμα μέλη, στην επόμενη ε, διάσκεψη κορυφής ε, θα πρέπει να στείλουμε αυτό το μήνυμα. Έχουμε τη δυνατότητα το 2014 να είναι μία καλή χρονιά πρέπει να υπάρξει ένα σκαρίφημα στην Επιτροπή για την Οικονομική Ένωση. Το πλαίσιο οικονομική διακυβέρνηση που έχουμε πλήρω εφαρμόσει για πρώτη χρονιά είναι ένα νέο εργαλείο και θα επιφέρει σημαντικέ βελτιώσει. Θα πρέπει όμως ε, να συμπληρωθεί. Θα πρέπει να καταβάλουμε περαιτέρω προσπάθειες ε, για να είναι σταθερή η περιοχή του ευρώ και τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι κάτι που οφείλουμε στους πολίτες μας, κάτι που οφείλουμε στις χώρες μας και ιδιαίτερα στις χώρες που κατέβαλαν τόσες προσπάθειες ε, για να ανακάμψουν μετά από μία κρίση. Θα πρέπει να προβλέψουμε την επόμενη κρίση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει πρωτίστως να ε, περατωθεί η Τραπεζική Ένωση, αλλά να υπάρξει και ένα νέο ταμείο. Η Επιτροπή εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες που καταβάλλονται για πρόοδο και η εφαρμογή των προτάσεων. Τώρα εναπόκειται στις χώρες μέλη να πάρουν μέρος σε αυτή τη συζήτηση και να καταλήξουν σε γενικές συμφωνίες. Κάποια πρόοδος επετεύχθη χθε στο Συμβούλιο και έχω τη βεβαιότητα ότι μία συμφωνία θα επιτευχθεί πριν από τη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου σε ό,τι αφορά τα νομοθετήματα αυτά πριν από τις εκλογές μετά από τη θεσινή συζήτηση έχουμε λόγους να θεωρούμε ότι θα υπάρξει συμφωνία για τις δύο προτάσεις που εκκρεμούν. Ελπίζουμε ότι οι αποφάσεις αυτές θα ληφθούν πριν από το τέλος του χρόνου. Η περάτωση της Τραπεζικής Ένωσης θα πρέπει να είναι ο πιο άμεσος στόχος μας. Παρόλα αυτά, αυτό είναι κάτι που ε, δεν, θα τελειώσει τόσο εύκολα. Θα χρειαζόμαστε περισσότερο αξιόπι, στα συστήματα για το συντονισμό των, των πολιτικών σε όλη την Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα θα συνεχίσει να εξετάζει τι συμβασιακέ σχέσει και του μηχανισμού αλληλεγγύη. Οι συμβασιακέ ρυθμίσει θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να εξασφαλίσουν τι σημαντικέ διαθροτικές μεταρρυθμίσει που θα πρέπει να γίνουν έγκαιρα. Αυτέ οι ρυθμίσει θα είναι ένα βήμα ακόμα που θα βελτιώσουν την κατάσταση στον χώρο μα και θα μας δώσουν τη δυνατότητα να δώσουμε οικονομικά κίνητρα για να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις. Η Επιτροπή υιοθέτησε μια ανακοίνωση σχετικά με αυτό στις αρχές του χρόνου. Θα ήθελα να πω για μία ακόμα φορά, αλλά αυτός δεν είναι ο ε, τρόπος για να δυσκολεύουν τα πράγματα οι Βρυξέλλες ε, ε, για τις χώρες μέλη. Αυτά ε, είναι θέματα τα οποία προβλέπονται στις συμφωνίες. Τώρα τίθεται το θέμα ενδυνάμωσης αυτής της συμφωνίας να μπορέσει να υπάρξει μεγαλύτερη εξέριξη, μεγαλύτερη συμμετοχή των συμφεροντούχων και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συμφωνηθεί. Θα πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα γίνουν πιο απτά, πιο συγκεκριμένα τα πράγματα για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις από τη στιγμή που είναι προς το κοινό συμφέρον όλων μας. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη δέσμευση προς όφελος ε, της ε, ε, ζώνης του ευρώ και όλης της Ευρώπης. Η Επιτροπή ελπίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα θέσει ορισμένες βασικές αρχές σχετικά με αυτά τα θέματα που θα αποτελέσουν την βάση για την περαιτέρω εργασία για το πρώτο ίμιση του 2014. Καταρχάς θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς σε ό,τι αφορά τις ε, ρυθμίσεις και τους μηχανισμούς αλληλεγγύης στο υπάρχον πλαίσιο του ε, εξάμεινου θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε, εκείνες, ε, σε εκείνους του τομείς που επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και θα πρέπει να συμφωνήσουμε και να εμπλέξουμε όλες τις χώρες σε ό,τι αφορά το θέμα του, της Νομιματικής Ένωσης θα πρέπει να υπάρξει στήριξη του προπολογισμού, εγγυήσεις ε, και θα πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις και δυνατότητα απορρόφησης των καραδασμών. Αγαπητά μέλη, το δεύτερο θέμα της, ε, της ημεσίας διάταξης είναι η κοινή ε, ασφάλεια. Θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή προσέγγιση στο θέμα της άμυνας. Τώρα περισσότερο από ποτέ η Επιτροπή λέει ότι θα πρέπει να επιτελεστεί πρόοδος και αυτό το επανέλαβε πάρα πολλές φορές ο πρόεδρος Μπαρόζο. Στην ανακοίνωση του προηγούμενου Ιουλίου σε ό,τι αφορά, που αφορούσε τον τομέα της άμυνας η Επιτροπή ε, τόνισε ακόμα περισσότερο το θέμα αυτό. Έχουμε διατυπώσει προτάσεις για μια λιγότερο κατακρεματισμένη αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη. Θέλουμε να υποστηρίξουμε και να δυναμώσουμε τις ε, στρατηγικές ικανότητες της Ευρώπης. Θα πρέπει να κινηθούμε προς ε, ένα ε, περισσότερο συνεκτικό τομέα της ασφάλειας καταρχάς, γιατί χρειαζόμαστε μια κοινή ορατή πολιτική που θα αποτελέσει απτή απόδειξη της δέσμευσης θα πρέπει να στηρίξουμε τις απόψει μα με συγκεκριμένε αποστολέ όταν καθίσατε κάτι τέτοιο αναγκαίο. Μέσω της γοργής ανάπτυξης των αποστολών μπορούμε να δείξουμε ότι πραγματικά τα καταφέρνουμε θα πρέπει να αποκτήσουμε τεχνογνωσία σε διάφορους ε, ε, τομείς. Θα πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις ε, στη διεθνή σκηνή. Δεύτερον, θα πρέπει να κινηθούμε ακόμα πιο πέρα στον ε, τομέα αυτό, γιατί υπάρχουν προβλήματα ε, που αφορούν τον τους προπολογισμού σε όλες τις, Ευρωπαϊκές τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, πάνω από το 75% των δαπανών στον τομέα της άμυνας δαπανώνται σε επίπεδο εθνικό. Δεν έχει νόημα ε, να χρειαζόμαστε 16 τύπους ε, πελικοπτέρων, θα μπορούσαμε να έχουμε μόνο ένα. Θα πρέπει να αναπτύξουμε κοινά ε, πρότυπα ε, ε, και να αναπτύξουμε την αυτονομία μας. Οι οικονομίες κλίμακας και θα πρέπει να ενδυναμώσει την στρατηγική μας ικανότητα. Σε αυτό το τομέα μιλάμε για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Ο τομέας αυτός απασχολεί 400.000 άτομα και δημιουργεί ακόμα περισσότερες ε, θέσεις εργασίας. Και όλοι μας γνωρίζουμε ότι έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κύκλο εργασιών. Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτές τις θέσεις εργασίας είναι απαραίτητο να υπάρχει ανταγωνιστικότητα ε, και καινοτομία. Θα πρέπει οι χώρες μας να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε νέα δίκτυα που ε, μπορούν να προωθήσουν τις πιο προηγουμένες τεχνολογίες στον τομέα της άμυνας. Οι χώρες μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν τις οδηγίες του 2009 σε ό,τι αφορά τις, ε, τις προμήθειες στον τομέα της έρευνας και θα πρέπει να ε, προωθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε σκοπό να κάνουμε περισσότερο για να μπορέσουμε να προωθήσουμε μια κοινή προσέγγιση στην πιστοποίηση και για να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών μας. Ε, ε αποδίδουμε πολύ μεγάλη ε, σημασία σε όλους τους τομείς που θα μπορούσαν να προωθήσουν τον τομέα της άμυνας. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ευρώπη. Η κοινή πολιτική ασφάλεια συνεπάγεται στενή συνεργασία με την ε, Αφρικανική Ένωση, με τα ε, ε, Ηνωμένα Έθνη. Και όλοι μαζί θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες εστιάζοντας σωστά τους στόχους μας. Συνεπώς, η συζήτηση, με τη συζήτηση αυτή που θα γίνει στο Συμβούλιο Επιτροπή ελπίζει να υπάρξει κινητήριο σε δύναμη για να πτυχθούν συνέργειε μεταξύ των χωρών μελών. Χρειαζόμαστε μια περισσότερο ανταγωνιστική και συνεκτική βιομηχανία. Αγαπητά μέλη, πάντοτε μας στηρίξατε μια πιο ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία βελτιώνει την ευημερία των πολιτών και παίζει καθοριστικό ρόλο στην διεθνή σκηνή. Θέματα επί των οποίων η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συνεργάστηκαν και συνεργάστηκαν απάντοτε τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία χρόνια ε, ε, συντελούν στην κινητήριο αυτή η δύναμη που οδηγεί στην πρόοδο. Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, η Επιτροπή θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα υποστηρίξει την ανάγκη να υπάρξουν συγκεκριμένες ε, δράσεις μέσω της Task Force για τη Μεσόγειο. Το, η περίπτωση της Λαμπεντούσα κατέστησε σαφές με έναν αλγινό τρόπο ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε περισσότερο στην περιοχή της Μεσογείου. Έδειξε τα όρια των εθνικών πολιτικών σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων όπως ε, παράνομες ροές μετανάστευσης. Έδειξε πόσο απαραίτητο είναι να στηρίξουμε χώρες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά την μετανάστευση. Θα πρέπει να δοθεί ε, ιδιαίτερη ε, στήριξη, ακόμα και έκταξη, έκτακτη στήριξη για την εποπτεία των ε, σύνορων. Η φύση των προβλημάτων απαιτεί μια τέτοια στήριξη, γιατί αυτό θα αποβεί προς όφερος όλων μας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, θα πρέπει να υπάρξει πρακτική συνεργασία και με τις τρίτες χώρες. τα ε, περιφερειακά προγράμματα θα μπορούσαν να γίνουν πιο ισχυρά, ιδιαίτερα για την Αφρική. Οι προσπάθειε μα θα, θα μπορούσαν να αποφέρουν περισσότερο και από κοινού με τι χώρε μέλη θα πρέπει να δούμε πώ θα μπορούσαν να, να ανοίξουμε νέε νομικέ οδού σε ό,τι αφορά τους ερευνητές ε, ή του φοιτητέ. Τέλο, θα πρέπει να αυξήσουμε τη συνεργασία μα με τις τρίτες χώρες. Ε, θα πρέπει να υπάρξει διάλογο για τη μετανάστευση, την ασφάλεια και αυτό θα πρέπει ε, να γίνει με την Αίγυπτο, τη Λιγία, την Αλγερία και το Λίβανο αξιότιμα μέλη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, λαμβάνει υπόψη την πρόοδο που έχει ε, καταγραφεί σε διάφορες προτάσεις. Ε, έχουμε να αναφέρουμε θετικά νέα, αλλά υπάρχουν ορισμένοι τομείς όπου χρειάζεται να επιτελεστεί πρόοδος. Οι χώρες μέλη θα πρέπει να τιμήσουν τις υποχρεώσεις τους. Για να σας παραθέσω ένα παράδειγμα, ε, η φορολογία και ιδιαίτερα η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Ένα πρόγραμμα δράσης υιοθετήθηκε πέρσι. Η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για ένα προηγμένο σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο φορολογικής ε, ε, διοίκησης. Ε, γίνονται διαπραγματεύσει με το Μόνακο, το Σαμαρίνο, την Ελβετία και το Λίχνεστάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασικό ε, παίκτη για τα παγκόσμια ε, πρότυπα. Για μία ακόμα φορά οι Υπουργοί Οικονομικών απέτυχαν να επιτύχουν συμφωνίε σχετικά με την οδηγία και τι για τις πωλήσει. Ε, θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πιέση στο πεδίο αυτό. Εν τέλει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ελπίζουμε ότι θα συμφωνήσει στο να δώσει σημαντική όθηση στη δυνατότητα για πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις τέτρα τις μικρομεσαίες. Έχουμε κάνει πρόοδο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ενισχύσει σημαντικά τις ε, δραστηριότητες της μετά τις συμφωνίες για τη διάθεση ε, χρηματοδότησης μέσω δικών της κεφαλαίων. Υπάρχουν ε, μέσα επιμερισμού κινδύνου τα οποία υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και επίσης υπάρχει πρόθεση να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο αυτές οι δραστηριότητες. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με μερικά σχόλια για την κατάσταση στην Ουκρανία. Ξέρω ότι έγινε συζήτηση στην Ολομέλεια εχθέ για την Ανατολική Γειτονία, εχθέ το απόγευμα. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε φυσικά να γνωρίσουμε στη σημερινή μα συζήτηση. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ιδιαίτερω και απερίφραστα τι θέσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ευρωπαϊκέ αξίε και αρχέ πρέπει να γίνονται σεβαστέ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερω για τι αρχέ τη Ουκρανία, όπω και για οποιονδήποτε άλλο βεβαίω. Ιδιαίτερω μετά τα όσα συνέβησαν εχθέ τη νύχτα, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και να επαναλάβουμε ότι ποτέ δεν είναι απάντηση η βία. Ε, η λύση πρέπει να βρεθεί με πολιτικά μέσα με το διάλογο με την ε, αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος Μπαρόσο έχει ήδη συνομιλήσει δύο φορές με τον πρόεδρο Γιαννούκοβιτς μετά την ε, διάσκεψη της Ρήγα, στο τηλεφωνικά του υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιείται βία για να κατασταλούν ειρηνικές διαδηλώσεις και να παραβιάζουν τα δικαιώματα των πολιτών. Η κάθε Άστον βρίσκεται και σήμερα στο Κίεβο επιτόπου για να συμβάλλει στην εξέβρεση μιας ειρηνικής λύσης και μια πολύ έντονη κατάσταση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ουκρανία. Ο λαός της Ουκρανίας έχει ξεκάθαρα διακηρύξει ότι υποστηρίζει την ευρωπαϊκή επιλογή της Ουκρανίας. Η προσφορά από πλευράς μας για την υπογραφή μιας συμφωνίας με την Ουκρανία για ένα ε, εις αλλά και εκτεταμένο χώρο ελεύθερων συναλλαγών παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρέπει βεβαίως να προχωρήσει το Συμβούλιο και με δεδομένες τις τωρινές εντάσεις ε, η επιλογή είναι μόνο μια ειρηνική λύση. Ε, ελπίζω ότι θα έχει αντίκτυπο και η ευρύτερη συνένεση που εκφράσατε και, χθες, και εσείς εχθές στην συζήτησή σας στο Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο θα συνεργαστούν προς το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σεύκοβιτς. Και τώρα εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο ο πρόεδρο Ιωσήφ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σχετικά με την Ουκρανία πρώτα απ' όλα. Παρακολουθούμε προσεκτικά το τι συμβαίνει εκεί. Ξέρουμε ότι δεν υπογράφηκε η συμφωνία αυτή και ο πληθυσμό της Ουκρανίας έχει βγει στους δρόμου για να υποστηρίξει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θέλω όμως να πω στους Ουκρανούς πολίτες ότι είμαστε στο πλευρό τους και ότι καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας εναντίον τους είναι σοβαρή κατάσταση, μπορεί να οδηγηθεί σε έκρηξη και γι' αυτό ζητάω στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο να υπάρξει διαμεσολάβηση όπως έγινε και με την Πορτοκαλή Επανάσταση για να βρεθεί μια δημοκρατική λύση. Οι Ουκρανοί πολίτες μας θέλουν ένα μήνυμα. Μας λένε ότι θέλουν μια ισχυρή Ευρώπη. Εξάλλου, και εντάξει, μάλλον χαίρομαι, είναι εκεί που βλέπουμε τις περισσότερες ευρωπαϊκές σημαίες, ενώ σε άλλες χώρες βλέπουμε όλο και λιγότερες. Οι φιλοδοξίες είναι μεγάλες και αν ε, βάλουμε τις βάσεις, ε, μια, πως βάλαμε μάλλον τις βάσεις για μια πραγματική οικονομική ένωση, αυτό είναι ήδη πολύ σημαντικό. Πριν από μερικά χρόνια κάτι τέτοιο θα ήταν ε, αδιανόητο. Ήταν καλές όμως αυτές οι αποφάσεις και τίποτα δεν χάσαν από την ταυτότητά τους οι χώρες μέλη. Η συμφωνία, οι έξι συμφωνίες μάλλον, οικονομικές συμφωνίες για τη διακυβέρνηση. Όλα αυτά είναι θετικά. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν και κάποια σημάδια διστακτικά μεν, αλλά υπάρχουν οικονομικές ανάκαμψεις. Άρα μαζί πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, είτε μας αρέσει είτε όχι. Εξάλλου δείτε τον οικονομικό τομέα. Τι γίνεται με τη συνεργασία. Ενώ οι πολιτικοί μερικές φορές θέλουν ο καθένας στη χώρα τους να δουλέψουν. Δεν είναι δυνατόν. Τα χρήματα δεν ε, είναι άπειρα. Γι' αυτό και χρειάζεται συνεργασία. Και εδώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριο Σεύκοβιτ και για την άμυνα. Μερικέ φορέ είναι δύσκολο, αλλά μερικέ χώρε χρησιμοποιούν λιγότερο από το 2% ε, του έπτους για την άμυνα. Αν λοιπόν δεν οργανωθεί η Ευρώπη και δεν προχωρήσουμε μαζί στην άμυνα, θα εξαφανιστούμε από την επόμενη τάξη του κόσμου. Ο κόσμος αλλάζει και μετά τον ψυχρό πόλεμο. Βλέπετε τι γίνεται στη Λιβύη, στη, στο Μαλί, στην Κεντρική Αφρική. Αν δείτε πώς θυσιάζονται αδύναμοι άνθρωποι στην Κεντρική Αφρική, μα εννοείται ότι η Ευρώπη έχει ρόλο και πρέπει να είναι εκεί παρούσα. Θα υπάρξουν όλο και περισσότερες αποστολές στις οποίες θα πρέπει να συμμετάσχει η Ευρώπη. Είναι δικιά μας ευθύνη, το δείχνουν αυτό οι καιροί. Και αν δεν το κάνουμε εμείς, ε, τι να γίνει, θα το κάνουν οι Ρώσοι στη θέση μας. Αρκεί να δούμε τι γίνεται δίπλα μας, στην Ουκρανία, στη Μολδαβία και κάποια από τα δικά μας στρατηγικά συμφέροντα μπορεί να απειληθούν από περιφερειακές δυνάμει. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι λοιπόν και το έχω ξαναπεί εδώ στο ημικύκλιο. Όχι για να πολεμήσουμε, για να κάνουμε πόλεμο, αλλά για να κρατήσουμε την ειρήνη, να προστατεύσουμε την ειρήνη. Τις βλέπετε τι εικόνε στην τηλεόραση και από την Κεντρική Αφρική. Στην επόμενη θητεία λοιπόν πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο για να ενισχύσουμε την κοινή μα πολιτική ασφάλεια και άμυνας αν θέλουμε να εξακολουθούμε να υπάρχουμε στον κόσμο, αλλά και για να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Αυτό σημαίνει να ενισχύσουμε την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε ακόμα και στρατιωτικά με μικτές δυνάμεις. Έχουμε κάποια αρχή με το Eurocorps, είναι μια αρχή μόνο. Έχουμε τις εννέα χώρες μέλη που συμμετέχουν στην κοινή ε, πολιτική μας, κάτι το οποίο όμως πρέπει να αλλάξει, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο. Και προσοχή, μην με παρεξηγήσετε, ε, συγχρόνως πρέπει να ενισχύσουμε και την ε, βοήθειά μας στην ανάπτυξη των ε, χωρών αυτών που βρίσκονται σε κρίση. Κεντρική Αφρική, για παράδειγμα, γιατί πραγματικά όταν χθε το βράδυ κοίταξα την τηλεόραση ήταν ένα σοκ για μένα. Δύο πράγματα χρειάζονται εκεί. Χρειάζεται η διατήρηση της τάξης για να αποφευθεί το δράμα και χρειάζεται και αναπτυξιακή βοήθεια που να αξίζει το όνομά τη όμως. Και επανέρχομαι γιατί κύριε Σεύκοβιτς είπατε αυτά που σκόπευα να πω εγώ. Πώς εξοπλίζουμε τι θετικές μα δυνάμει, και αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να βάλουμε από κοινού του πόρου μα για έρευνα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να δουλεύουμε όπως κάναμε μέχρι τώρα ο καθένα μόνο του. Το είπατε, να δούμε τα διάφορα υλικά. Εγώ δεν είμαι ειδικό για τα υλικά, αλλά προφανώ και πρέπει να συνεργαστούμε και με τον ΝΑΤΟ για να μπορέσουμε και εκεί να έχουμε μια αμυντική βιομηχανία που να αξίζει το όνομά τη και να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει στην Ευρώπη, να είναι βιώσιμη. Έχουμε τεχνολογία, έχουμε άμυνα, πρέπει να την απτύξουμε περισσότερο για να μπορέσουμε να κρατηθούμε στη θέση μας και να αντιμετωπίσουμε και την οικονομική κρίση. Το six-pack για την άμυνα, μια που είναι πολύ της μόδας ε, αυτός ο όρος, πρέπει να υπάρχει με στόχους που να μην είναι ταμπού. Το ζήτημα, συνάδελφοι, που τίθεται σήμερα όταν βλέπουμε τις εξελίξεις, που εντάξει μετά από κάθε επανάσταση υπάρχει εξέλιξη, revolution, evolution. Το είπανε και ορισμένοι συνάδελφοι και το six-pack για την δικαιοσύνη, για το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Δύσκολος φάκελος και αυτός. Δεν λέω ότι πρέπει να υποστηρίζουμε εμεί τον χ ή τον ψ, όχι. Αλλά υπάρχει μια λειτουργία της δικαιοσύνης που μας έλειψε. Δηλαδή μπήκαν διάφορες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες όμως δεν είχαν ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις τους πλήρως. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός αυτό, άρα η Ευρώπη πρέπει να δράσει και στον τομέα αυτό. Μην το ξεχνάμε όταν βλέπουμε τι γίνεται στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ευρώπη είναι μια κοινότητα αξιών, κοινών ευθυνών. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να ενισχυθεί για να έχει τη θέση της στη νέα τάξη στον κόσμο. Και όσοι θέλουν λιγότερη Ευρώπη, εγώ λέω όχι. Μεθαύριο χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Γιατί αυτοί που λένε ότι χρειαζόμαστε λιγότερη Ευρώπη σφάλουν και θα το διαπιστώσουν πολύ γρήγορα. Πρέπει να υποστηρίξουμε τι αξίε μα, τι κοινέ μα αξίε και να προχωρήσουμε, να πάμε μπροστά για το μέλλον και την κυριαρχία τη υπήρου μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα, εκ μέρου τη Ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο Πρόεδρο τη, κύριο Βόμποντα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω και εγώ με την Ουκρανία. Βεβαίως, θα πρέπει να καλέσουμε όλες τις δυνάμεις στη χώρα να περιορίσουν τις δράσεις τους, δραστηριότητες τους και να μην μεταρχόνται βία. Είναι καλό το ότι ο κύριος Γιαννούκοβιτς συνάντησε την κάθε άστον και τους πρώην προέδρους αλλά δεν αρκεί αυτό. Δεν αρκεί δηλαδή να κάθεται σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων να μιλάει με αυτού του ανθρώπου και από την άλλη πλευρά η αστυνομία να καταστέλει βία τι διαδηλώσει. Εμεί πρέπει να σταθούμε στο πλευρό των ανθρώπων που αγωνίζονται και διαδηλώνουν στην ε, Ουκρανία για την Ευρώπη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί γι' αυτό αγωνίζονται. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι όντω σωστό ότι χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για την άμυνα, για να αναφερθώ στο θέμα αυτό, στην άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν προβλήματα σε διάφορες περιοχές και όχι τόσο στην Ευρώπη. Πρέπει όμως να αναλάβουμε εμεί τα καθήκον μας, δεν μπορούμε να είμαστε οι παλιά και λησμονημένη Ήπειρος, πρέπει να αναλάβουμε δράση, φερρυπίν κατά της τρομοκρατίας. Ε, μία πληγή που μας μαστίζει εδώ και πολύ καιρό. Ε, έγινε λόγος για συνεργατικές δράσεις, για ε, συγκέντρωση πόρων και συνδυασμό πόρων στην άμυνα Βεβαίω, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και να ενισχύσουμε τι προσπάθειέ μα για την άμυνα. Εάν τώρα μάλιστα κινδυνεύουν με, από την EADS 6.000 θέσει εργασία, αυτό οφείλεται στο ότι δεν συνεργάζονται οι κυβερνήσει των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ενισχύουν, δεν υποστηρίζουν τι ευρωπαϊκέ αμυντικέ δομέ και τι ευρωπαϊκέ αμυντικέ βιομηχανίε. Χρειάζεται, γι' αυτό είναι ένα σκάνδαλο. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε περισσότερε προσπάθειε. Χρειάζεται όμω ταυτόχρονα και κοινωνική συνοχή και οικονομική ανάπτυξη για να εξασφαλίσουμε την υποστήριξη του Ευρωπαίου πολίτη. Και έτσι περνώ στην οικονομική κατάσταση. Ναι, ακούσαμε υπέροχα νέα τις τελευταίες ημέρες. Ε, κτιμόμενη ετήσια ανάπτυξη που αναθεωρήθηκε από το 2,8% στο 3,6%. Με μείωση της ανεργίας από το 7,3% στο 7%. Με τα χαμηλότερα ποσοστά από το Νοέμβριο του 2008. Τέλεια, πολύ ωραία νέα. Μόνο που αυτά είναι τα στοιχεία για τις ΗΠΑ και όχι για την Ευρώπη. Στην Ευρώπη δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα όπω μα τα περιέγραψε το Συμβούλιο και η Επιτροπή σήμερα. Έχουμε πολλέ δυσκολίε ακόμη και έχουμε δείξει ότι μπορούμε με μια ανεξάρτητη δράση να έχουμε και διαφορετικά αποτελέσματα αλλά δυστυχώ δεν αλλάζει στάση και πολιτική επιτροπή ούτε και πολύ μέσα στο Συμβούλιο. Και γι' αυτό θα πρέπει να πω Έχοντα επισκεφθεί αρκετέ χώρε που αντιμετωπίζουν κρίση, όσο πιο πολύ ανοίγει το στόμα του ο κύριος Ρέν, όσο πιο πολλές συνεντεύξει δίνει, τόσο ενισχύονται τα αντιευρωπαϊκά συναισθήματα στις χώρες αυτές. Εγώ δεν θέλω να να ε, παρεμβληθώ στο διαγωνισμό ομορφιάς μεταξύ Φερχόφστατ και Ρεν. Δική τους δουλειά είναι. Αλλά πρέπει να αλλάξουν πολιτική. Εδώ έχουμε να κάνουμε με 18% σωρευτική ε, απώλεια ε, παραγωγικότητας για την Ελλάδα, 19% για την Ισπανία και τη Γαλλία. Και ο κύριος Ρεν μας λέει, η Επιτροπή και το Συμβούλιο, ότι η Ισπανία θα έχει το 2033 φτάσει στο μέσο όρο ανεργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να κοιτάμε μόνο τα όρια, να λέμε και τα υπόλοιπα. Πώς λοιπόν μπορούμε να ζήσουμε από την Ελλάδα στην Πορτογαλία. Πώς μπορούμε να δούμε, γιατί βλέπουμε ότι ανεξάρτητοι οργανισμοί, όχι οι συγκεκριμένε πολιτικέ δυνάμει, καταγράφουν αυτή τη ε, δυσφορία. Όταν η Τρόικα στην Ελλάδα λέει Α, βγάλτε από τα σπίτια του ανθρώπου, υπάρχουν και άστεγοι. Αν δεν μπορούν να πληρώσουν το νίκη του ή το, το δάνειό του. Και τι απάντηση δόθηκε από κάποιον ε, από τους Τροϊκανούς, φτιάχτε τους ε, στέγες αστέγων. Άμυνο άστεγε, προσφέρετε τους άσυλα. Αυτό είναι η απάντηση που δίνει η Τρόικα σε ορισμένες χώρες και βέβαια δεν βοηθάει καθόλου. Ούτε το δεχόμαστε εμείς αυτό. Επίσης δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα του 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ που προσφέρεται στις τράπεζες για ε, ε, που ορίστηκε ως πρόστιμο για τράπεζες. Γιατί αυτό να μην πάει λοιπόν στην ανεργία, γιατί να μην χρηματοδοτήσει τον αγώνα για την καταπολέμηση ανεργίας και για την εξασφάλιση μιας καλύτερης ευκαιρίας για τους νέους. Και μπορώ να ε, πω ότι αυτά είναι πολύ πιο σημαντικά από τι συμβατικέ συμφωνίε που αναφέρατε, κύριε, Πρόεδρε, κύριε εκπρόσωπε της Επιτροπής και από όλα τα ζητήματα τα οποία ε, αφορούν την ε, λειτουργία τη Οικονομική και Νομισματικής Ένωση, γιατί πρέπει να στερθούμε περισσότερο στον κοινοβουλευτισμό. Επιτρέψτε μου λοιπόν να αναφερθώ σε κάποιε συγκεκριμένε πτυχέ τη κατάσταση στην Ευρώπη σήμερα. Πριν από 40 και, και χρόνια, 40 χρόνια ακριβώ στι 13 Νοεμβρίου, για να είμαι ακριβή, 40 χρόνια λοιπόν πριν, μίλησε ο Γερμανό καγκελάριο Βίλι Μπραντ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με μία ομιλία ενός μεγάλου οραματιστή όπου μίλησε για μια κοινωνική Ευρώπη, για κοινωνικά δικαιώματα, για οικονομική ανάπτυξη. Και εμείς βρισκόμαστε σήμερα, 40 χρόνια μετά, να αγωνιζόμαστε πάλι σε μια διελκυστήντα με την Επιτροπή και την πλειονοψηφία του Συμβουλίου για να ζητούμε περισσότερα κοινωνικά δικαιώματα, για περισσότερα και εντονότερα κοινωνικά κριτήρια στην ΟΝΕ. Αντί όμως να χτίζουν μια κοινωνική Ευρώπη, ορισμένες κυβερνήσεις στο Συμβούλιο και κοιτάω προς την Βρετανική κυβέρνηση, αλλά δεν είναι μόνο αυτή, προσπαθούν να ανοίξουν νέα χάσματα και διχασμούς και λένε ότι Φερρυπίν στα δικά του σύνορα, τα δικά του σύνορα μπορεί να τα περάσει κανείς μόνο αν έχει υψηλά εισοδήματα. Αντί να καταπολεμούμε λοιπόν τη φτώχεια, καταπολεμούμε, πολεμάμε κατά των πολιτών των άλλων κρατών μελών. Οι εθνικισμοί λοιπόν επικρατούν των κοινωνικών μελημάτων. Και αντί να δημιουργούμε θέσει εργασία για του πάντε και να καλύπτουμε το χάσμα μεταξύ φτωχών και πλουσίων, αντί να εξασφαλίσουμε καλύτερη κατανομή του παραγόμενου κέρδου, έχουμε αρχίσει να μιλάμε για ημεδαπού και αλλοδαπού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλοδαπού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε ήταν η Βρετανία είτε άλλα κράτη-μέλη ζητούν περισσότερα δικαιώματα και ισχύ που θα έπρεπε αντίθετα αυτά τα δικαιώματα ή την ισχύ της εξουσίας που έχουν να τα αξιοποιούν για να ελέγξουν εάν υπάρχει κάποιο τύπος, ε, τύπου τουρισμός ε, κοινωνικών επιδομάτων ας τον καταπολεμήσουν και θα τους βοηθήσει και η Επιτροπή με τα στοιχεία που έχει αλλά όχι περιστέλλοντας την ελευθερία της διακίνησης γιατί δημιουργείται μια διαφορετική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ένας λέει ας περιοριστούμε μόνο στην οικονομική αγορά ή στην αγορά για τις υπηρεσίες, στην κοινή αγορά φερρυπίν έστω και για τα αμυντικά προϊόντα. Αλλά υπάρχει και άλλο όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό περιλαμβάνεται και η ελευθερία για την εργασία και για τη διακίνηση και κατάσταση σε άλλη χώρα. Υπάρχει και άλλο όραμα για την Ευρώπη που λέει καταπολεμάμε την φτώχεια, που λέει καταπολεμάμε το όλο και ενισχυόμενο χάσμα μεταξύ εισοδημάτων των πολιτών. Δυσπιστία υπάρχει εναντίον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό οφείλεται στο ότι δεν δίνει λύσει στα προβλήματα, τα κοινωνικά και οικονομικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν είχαμε μια σαφέστερη οικονομική πολιτική, μια ισχυρότερη οικονομική πολιτική και κοινωνική ένωση, τότε θα μπορούσε η Ένωση και να ενισχύει την ελευθερία και την ελευθερία εργασία. Α μην καταστρέψουμε λοιπόν την Ευρώπη, α την ενισχύσουμε και α χτίσουμε την κοινωνική Ευρώπη ω βάση εμπιστοσύνη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα εκ μέρους της ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων, ε, ο κύριος Φερχόφστατ. Ευχαριστώ. Θέλω πρώτα απ' όλα να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Σβόπεδα για τις ελευθερίες που έχουμε. Μα για, σε εμά τους φιλελεύθερους υπάρχει η δημοκρατική επιλογή. Εμείς την υποστηρίζουμε. Είναι προφανές. Πέραν αυτού όμως θέλω να αρχίσω, Πρόεδρε, με φόρο τιμής απέναντι στους πολίτες της Ουκρανίας. Και γιατί? Γιατί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που έχουν βγει στους δρόμους του Κιέβου, κατά τη γνώμη μου, σήμερα είναι η καλύτερη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε στους ε, σκεπτικιστές απέναντι στην Ευρώπη. Γιατί με εθνικισμό και λαϊκισμό ορισμένοι προσπαθούν να πούνε ότι τελείωσε η Ευρώπη, ότι δεν υπάρχει μέλλον για την Ευρώπη. Όμω βλέπετε εκτός Ευρώπης, στου δρόμους του Κιέβου, ότι ένας άνθρωποι θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελπίδα μου λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι είναι ότι αυτό το πνεύμα υπέρ της Ευρώπης δεν θα κυριαρχήσει μόνο στους δρόμους του Κιέβου την επόμενη εβδομάδα αλλά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Και αυτό γιατί δεν πρόκειται για ένα κοινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπάρχουν τρία πολύ σημαντικά ζητήματα που πρέπει να ξεπεράσουμε την επόμενη εβδομάδα, έξι μήνες πριν από τις ευρωεκλογές. Το πρώτο είναι η Ευρωπαϊκή Άμυνα. Αμα ακριβώς πριν από 60 χρόνια, αγαπητοί συνάδελφοι, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση, κατά τη γνώμη μου, έπραξε ένα σοβαρό σφάλμα. Θα το θυμόσαστε. Το 54 ήταν, Μόλις είχα γεννηθεί πριν από ένα χρόνο. Δεν το θυμάμαι. Αλλά ξέρω ότι τότε η Γαλλική Εθνοσυνέλευση αρνήθηκε την ε, κοινότητα άμυνας, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άμυνας. Σφάλμα λοιπόν. Σήμερα και η κοινή γνώμη είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Υπάρχει πλειοψηφία, ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν υπάρχει ένα θέμα στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, που πρέπει να κάνουμε μαζί, αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Άμυνα. Και πριν από 10 χρόνια ξέρω ότι γελούσαν ε, μικροί όταν με τη, μερικοί όταν με τη Γαλλία και τη Γερμανία πριν από 10 χρόνια μετά δηλαδή από τον πόλεμο στο Ιράκ είχαμε πει ότι πρέπει να στηριχτούμε στις συμφωνίες σαν μαλό ανάμεσα στην Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και να φτιάξουμε την Ευρωπαϊκή Άμυνα, γελούσαν λοιπόν μερικοί. Δέκα χρόνια μετά η ιδέα αυτή μπορεί και πάλι να ανθίσει. Γιατί από πλευράς λιτότητας όλες οι χώρες μέλη αντιμετωπίζουμε δυσκολίες δημοσιονομικές. Οπότε δεν είναι πολυτέλεια πια η συνεργασία αυτή. Δεν είναι δυνατόν μάλλον να επιτρέψουν σε αυτού μα αυτή την πολυτέλεια ο καθένα μόνο του 28 χώρε να προχωρούν σε αυτόν τον τομέα. Όχι, πρέπει να συνεργαστούμε μαζί. Και υπάρχουν και άλλα θέματα. Υπάρχει οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό είναι το δεύτερο για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Κύριε Επίτροπε, εσεί εδώ ε, στηρίξατε τι βασικέ ρυθμίσει που όμω δεν θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή την ιδέα ότι ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη πρέπει να υπάρχει μια σύμβαση για μια συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, είτε πρόκειται για εργασιακή είτε κάτι άλλο και να υποβάλλεται μια τέτοια. Όχι, τότε έχουμε το θάνατο της Ευρώπης αν προχωρήσουμε με αυτές τις συμβασιακές ρυθμίσεις, γιατί θα υπάρξει αντίσταση σε όλες τις χώρες μέλη. Διότι ο κόσμος θα τις δει σαν ανάμειξη της Ευρώπης σε μια συγκεκριμένη εθνική μεταρρύθμιση. Το έχουμε ήδη πει και ο κύριο Μπρόκ και εγώ και ο κύριο Γκαλτιέρη εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το έχουμε πει στι διάφορε επιτροπέ. Και εσεί τι κάνετε, συνεχίζετε. Με Επιτροπή πρέπει να βρει μια άλλη ιδέα. Μια που να υποστηρίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύγκληση. Πρέπει να, υπάρχει, να υπάρξουν οδηγίε σύγκληση που να εφαρμόζονται και στι 28 χώρε μέλη και στι 17 χώρε τη Ευρωζώνης. Και αυτές οι κατευθυντήριε γραμμές σύγκλησης θα έχουν βέβαια διαφορετικές συνέπειες στη μία και στην άλλη χώρα με διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, εντάξει. Αλλά σταματήστε επιτέλους με αυτή την ιδέα των συμβασιακών ε, ρυθμίσεων, γιατί δίνουν την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πραγματικότητα αναμειγνύεται και επιβάλλει μια συγκεκριμένη εθνική μεταρρύθμιση, ενώ την ευθύνη κανονικά έχουν τα κράτη-μέλη. Τέλος, Πρόεδρε το τρίτο μου σημείο, η Τραπεζική Ένωση. Πρώτα απ' όλα, και το έχω επαναλάβει πολλές φορές εδώ στην Ολομέλεια, νομίζω ότι χωρίς την Τραπεζική Ένωση δεν υπάρχει λύση στην κρίση. Διότι θα καταλήξουμε σε αυτό που είχε και η Ιαπωνία. Δηλαδή ε, θα υπάρξει στασιμότητα. Υπάρχει το θέμα της χαλαρής, του χαλαρού συντονισμού. Αυτό δεν θα λειτουργήσει. Εμείς δεν θέλουμε διακυβερνητικό σύστημα, θέλουμε κοινοτικό σύστημα. Και διάβαζα και σήμερα το πρωί ποιο είναι το αποτέλεσμα του Συμβουλίου Κοφίν χθε το βράδυ. Διακυβερνητικό σύστημα. Κάτι το οποίο εμείς δεν θα δεχτούμε ποτέ. Ελπίζω. Και τέλο, στήριξη στου φορολογούμενους. Δεν πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι αυτοί που πληρώνουν την ύφη, οι τράπεζε. Γιατί και πάλι, αν είναι ένα σύστημα σαν και αυτό που είχαμε κατά το παρελθόν, πάλι την ύφη θα την πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Όχι, οι τράπεζε πρέπει να πληρώνουν ανάλογα με το προφίλ του. Πρόεδρε, ελπίζω όλοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσουμε να στηρίξουμε πλήρω την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να ανταποκρίνεται σε αυτό. Αν κατακλείδη, ελπίζω ότι το Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα και το κοφίν θα έχουν το ίδιο ευρωπαϊκό πνεύμα σαν και αυτό που έχουμε σήμερα στο Κίεβο και στην Πλατεία Ελευθερίας εκεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φερχόφστατ. Ο Σαλφός Οντί έχει μια ερώτηση να σας απευθύνει. Παρακαλώ κύριε Οντί. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, αναφερθήκατε στους ε, Γάλλους βουλευτές που πολύ σωστά προτίμησαν να μην αναμίξουν την άμυνα με την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, γιατί δεν ήταν έτοιμη τότε η Ευρώπη. Ερωτώ λοιπόν, εσείς πιστεύετε ότι η Ευρώπη σήμερα είναι σε θέση να αναλάβει την άμυνα των λαών? Μπορείτε να εξασφαλίσετε τη λειτουργία της άμυνας χωρίς τα μεγαλύτερα κράτη, αυτά που είναι σε θέση να έχουν και τους μεγαλύτερους στρατούς. Είναι πράγματι η Ευρώπη έτοιμη σήμερα. Απάντηση. Νομίζω, κύριε Οντή, καταρχάς, ότι η Ευρωπαϊκή Άμυνα πρέπει να προχωρήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν αρκεί μόνο μία χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχουμε αρκετά μέσα οικονομικά για να καλύψουμε τις δαπάνες της. Τα ευρωπαϊκά ε, κράτη δαπανούν 42% των, του ύψους των δαπανών των ΗΠΑ. Τεράστιο ποσό γιατί οι ΗΠΑ έχουν τις μεγαλύτερες δαπάνες. Με αυτό όμως το ποσό, το 42% το τεράστιο, μόνο 10% σε αναλογία με τις δράσεις των Αμερικανών μπορούμε να αναλάβουμε. Δηλαδή είμαστε 4 με 5 φορές, αν κάνει κανείς τον υπολογισμό, 4 με 5 φορές λιγότερο αποτελεσματικοί από τους Αμερικανούς στον χώρο της άμυνας. Άρα λοιπόν ναι, πρέπει να χτίσουμε πάνω του μαλό τη συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Μεγάλης Βρετανίας για να ξεκινήσει η κοινότητα άμυνας. Και εγώ προτείνω με εκείνη την ε, σύνοδο με τον κύριο Σιράκο που ήμουν παρόν πριν από 10 χρόνια που ανέφερα νωρίτερα όπου είπε ότι πρέπει πλέον να προχωρήσουμε, να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό ο κύριος Πρόεδρος. Κύριε Φερχόφιστα, ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Χάμς εξ των Πρασίνων. Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι τώρα πια που οι ειδικές δυνάμεις αστυνομίας έχουν ε, οι ειδικέ δυνάμει ασφαλεία έχουν ε, εκενώσει τα γραφεία των, ε, του κόμματο αντιπολίτευση που έχει καθαρίσει αυτή η κατάσταση στην, ε, στο Κίεβο. Μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε σε σαφεί καταδίκε. Λυπάμαι που δεν υπήρχε τέτοια βούλη στο προηγούμενο, την προηγούμενη εβδομάδα, που δεν υπήρχε κάποιο εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να τοποθετηθεί εγκαίρω, που ίσω θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει αυτέ τι εξελίξει. Το ψήφισμα το οποίο χθε συζητήσαμε και θα ψηφίσουμε σήμερα έπρεπε να έχει έρθει πιο νωρί. Επιδεικνύεται λοιπόν στην περίπτωση αυτή του Κιέβου ε, μεγάλη αδυναμία από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αδυναμία να προχωρήσει με μια ενιαία πολιτική και να αναλάβει πραγματική δράση. Για την Ουκρανία το πρόβλημα αυτό τονίζεται ιδιαίτερα και αφορά ουσιαστικά την αδυναμία μας να κάνουμε ενωμένα μία πολιτική έναντι της Ρωσίας. Οι Ουκρανοί, οι Ουκρανίδες τώρα υποφέρουν λόγω αυτής της αδυναμίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα κληθούν να πληρώσουν τα σπασμένα. Για την ε, κοινή πολιτική άμυνας. Έχουμε εδώ ένα κίνδυνο να προσπαθήσουμε να ε, ζεύξουμε το άλογο από τα οπίστια του και όχι από, από τα, να προσπαθήσουμε τραβήξουμε το άλογο από τα οπίστια του και όχι από τα μπρος. Ας μάθουμε λοιπόν τι έχουμε κάνει από την Αταλάντα, από τη γαλλική παρέμβαση στο Μαλί, από τις κοινέ δράσεις, από την ε, εκένωση Ευρωπαίων ε, στρατιωτών εντό εισαγωγικών από το Αφγανιστάν, ε, η διαφυγή καλύτερα. Τι μαθαίνουμε ότι χρειάζεται μια καλύτερη και κοινή πολιτική δεδομένου ότι είναι περιορισμένα τα μέσα, τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η κατάσταση ε, είναι τέτοια που δίνουμε πολύ λίγα ελάχιστα για την κοινή κοινωνική πολιτική, για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν δίνουμε σε αυτόν τον προϋπολογισμό αρκετά ε, ποσά. Τώρα το να λέμε ότι θα δώσουμε πιο πολλά για την άμυνα δεν καταλαβαίνω που έχουμε φτάσει. Είναι δυνατόν αυτό να είναι η, ε, το πνεύμα που ε, διαπνέει την Ευρωπαϊκή Ένωση. για δε τη συνεργασία μεταξύ των οργάνων, χωρί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και το έχουμε συστήσει χιλιάδε φορέ, χωρί το Σβεν Κίνγκολτ, χωρί τον ε, Φιλίπ Λάμπερτς δεν θα είχαμε καν τον πρώτο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης ούτε την εποπτεία των τραπεζών. Για να μιλήσουμε δε για την δικαιοσύνη κύριε Σεύκοβιτς στην Ευρώπη το ταμείο αυτό στήριξη το οποίο έχουν εξασφαλίσει προς όφελός τους οι τράπεζες είναι για μένα μία ενευκό επιταγή, γιατί χωρίς αυτό δεν προχωρεί τίποτα. Ο κύριος Φερχόφστατ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέρθηκε στις προκλήσεις ε, την ανάγκη να εξασφαλίσουμε τα μέτρα εκείνα που θα ε, σταθεροποιήσουν ακροπρόθεσμα το ευρώ για μια κοινή φορολογική και οικονομική πολιτική. Αυτό όμως το οποίο μας προτείνετε εσείς κύριε Σεύκοβιτς είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι το αντίθετο. Ποιος θέλει να επαναληφθεί αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Μία χώρα η οποία στην αρχή όλης αυτής της συζήτησης ήταν διατεθειμένη να συζητήσει για μεταρρυθμίσεις, όπου υπήρχε θετικό κλίμα υπέρ των μεταρρυθμίσεων και να βρίσκεται τώρα σε αυτήν την κατάσταση κατά την οποία οι μεταρρυθμίσεις επιβάλλονται μόνο και μόνο από το φόβο της επιβίωσης και όπου όλο και ενισχύονται τα ακραία ε, εθνικιστικά και δεξιά κινήματα γιατί πια δεν υπάρχει ελπίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ποιος θέλει να εξυπηρετήσει αυτήν την προοπτική με τις λεγόμενες συμβατικές σχέσεις όπως μας τις παρουσιάζετε εσείς. Ποτέ δεν πρόκειται να συμφωνήσει η ομάδα μου σε αυτό κύριε Σεύκοβιτς. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Χάρμς. Εκ μέρους των συντηρητικών ο κύριος Κάλαναν. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλήσαμε πάρα πολλέ φορέ για το θέμα τη οικονομική πολιτική. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο θέμα τη αμυντική πολιτική. Όταν τίθεται το θέμα τη αμυντική πολιτική στην Ευρώπη, μία σωστή προσέγγιση θα πρέπει να αφορά συμβατότητα, ικανότητα και συνεργασία. Και αυτή είναι η προσέγγιση που έχει υιοθετήσει η Ευρώπη εδώ και 60 χρόνια υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι μία δοκιμασμένη ε, συμμαχία, μολονότι πολλοί προσπαθούν να την υπονομεύσουν μέσω της γραφειοκρατίας. Αυτό ε, σημαίνει ότι προσπαθεί να ε, δημιουργηθεί από την πίσω πόρτα ένα ευρωπαϊκό στρατό. Όλοι αναγνωρίζετε ότι θα πρέπει να εξυγχρονιστεί το ΝΑΤΟ. Όταν έγινε το 49 για πρώτη φορά, ο πρώτο γενικό γραμματέα του είπε ότι ο ρόλο του ήταν να κρατηθούν οι Ρώσοι εκτό, οι Αμερικανοί εντό και οι Γερμανοί κάτω. Ε, βέβαια, τα πράγματα έχουν ανάξει από το 49. Η δύναμη της Ατλαντικής Συμμαχίας έγκυται στην σχέση, την Ατλαντική σχέση που περιέχει. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να κρατήσουμε τους Αμερικανούς εντός. Η Αμερικανική και η Ευρωπαϊκή συνεργασία είναι περισσότερο σημαντική από ποτέ. Δυστυχώς, υπό τον πρόεδρο Ομπάμα, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε διατρέχουν τον κίνδυνο να εστιάσουν την προσοχή τους στις δυτικέ ακτές. Εμείς τους πρόχνουμε, τους διώχνουμε. Ορισμένοι λένε ότι η μοναδική λύση είναι μια κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Ε, Τέτοιο όμω στηρίζεται σε πολλά επίπεδα. Καταρχά, οι ευρωπαϊκέ χώρε δεν έχουν του απαραίτητους απαιτούμενου πόρου. Το ΝΑΤΟ <clears throat> δαπανά ένα τρίσεκατομμύριο εκατομμύριο δολάρια για την άμυνα. Δύο τρίτα προέρχεται από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Το ένα τρίτο δαπανάται ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 75% από τέσσερι ευρωπαϊκέ χώρε. Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία αυτή δεν είναι ευρωπαϊκή άμυνα από τη στιγμή που τόσο λίγες χώρες σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος. Εάν προσθέσουμε τη συνολική ευρωπαϊκή δαπάνη, καταλαβαίνετε ότι χρειά μπροστά στη δαπάνη των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεύτερον, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν πρόκειται να δώσουν τον έλεγχο στη ε, ε, στρατηγία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, ε, ε, Βεβαίω αυτό είναι εκτός, ε, <clears throat> δεν τίθεται καν. Συνεπώ, υπάρχουν διακυβερνητικέ συμφωνίε συνεργασία των χωρών και ανάληψη δέσμευση. Κατά την άποψή μου, μου θυμίζει το ΝΑΤΟ. Αυτή είναι μια επικάλυψη. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι πόροι που ήδη είναι περιορισμένοι. Αυτοί είναι πόροι που θα μπορούσαμε να δαπανίσουμε στον τομέα της κατάρτισης και των εξοπλισμών αντί να παίζουμε με τα στρατι... Ε, ε, στρατιωτάκια. Το θέμα αφορά τα ίδια τα στρατεύματα. Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας έχουμε απόλυτο σεβασμό για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας και θέλω να αποτίσω φόρο τιμής για όσους ε, έχουν θυσιαστεί οι άνθρωποι αυτοί αντιπροσωπεύουν ε, τη χώρα μας, τη χώρα σας. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν την επιθυμία να πολεμήσουν και ενδεχομένω ε, να θυσιαστούν για, την, ε, για τα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Δεν είμαι σίγουρος όμως οι ευρωπαϊκές χώρες ήδη έχουν μια μακρά ιστορία διμερών και πολυμερών σχέσεων συνεργασίας. Και βεβαίως αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον βεβαίως θα πρέπει να συνεργαστούμε όπου κάτι τέτοιο είναι δυνατόν. τα προβλήματα θα ξεπεραστούν μέσα από αυτή την προσέγγιση. Βεβαίως αυτό αποτελεί και μέρος της πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ. Στην πρόσφατη αποστολή στο Μαλί χρησιμοποιήθηκαν ευρωπαϊκά ε, αεροπλάνα παράλληλα με αεροπλάνα βρετανικά. Αυτό είναι το είδος των μέτρων που δεν χρειάζονται μια νέα γραφειοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Απλά και μόνο χρειάζεται η βούληση των χωρών. Ε, δεν δεν πάντοτε την ίδια τάσεις σε όλες τις χώρες μέλη. Ας μην ξεχνάμε το πόσο μας χώρισε ο πόλεμο του Ιράκ πριν από 10 ε, χρόνια. Μα έδειξε απόλυτα καθαρά ότι η εθνική ανεξαρτησία είναι καθοριστική για πολλέ χώρε. Σε αυτού τους δύσκολου καιρού. δεν έχουμε την πολυτέλεια δύο αμυντικών οργανισμών στι Βρυξέλλε. Έχουμε έναν επιτυχή οργανισμό, υφίσταται ε, εδώ και 60 χρόνια, ε, και συνεχίζει να εκπροσωπεί την ελπίδα μας για την ασφάλεια του 21ου αιώνα. Κάθε βήμα που υιοθετούμε για μια κοινή ευρωπαϊκή ε, άμυνα μας απομακρύνει από το ΝΑΤΟ. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, δεν θα, πρέπει να επαγρυπνούμε και να είμαστε πάντοτε ενωμένοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μάθει από την κρίση, θα πρέπει να ε, μην ε, βιαζόμαστε, θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας πρακτικά σε αυτά που είναι λειτουργικά, όχι να δημιουργούμε νέες, νέους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς. Το, το ΝΑΤΟ είναι λειτουργικό. Ας παραμείνουμε εδώ και ας μην προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε στα παρασκήνια ένα ευρωπαϊκό στρατό και ας κοιτάξουμε να αυξήσουμε τη συνεργασία μας και την ε, ε, συμβατότητα. Σας ευχαριστώ από την Ενωτική Αριστερά η Πρόεδρος κυρία Τσίμερ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Εχθές ε, η οργάνωση για την απαγόρευση των χημικών όπλων ε, τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Πέρσι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί λοιπόν να μην αξιοποιηθεί η Σύνοδο Κορυφή τη προσεκού εβδομάδα ώστε να ε, προβληθεί ένα πραγματικό όραμα, ένα όραμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ένωση εκείνη η οποία πρόκειται να συμβάλλει το μέγιστο στην απαλλαγή του κόσμου σε διεθνές επίπεδο από τα χημικά όπλα, από τα όπλα μαζικής καταστροφής. Το 80% των χημικών όπλων ανά τον κόσμο έχει καταφέρει να, από, να ε, καταστρέψει αυτός ο οργανισμός ε, για την καταστροφή των χημικών όπλων. Τώρα προχωρήστε μια πολύ δύσκολη αποστολή και εμείς τι κάνουμε, οργανώνουμε μια συνοδοκορυφή για τους εξοπλισμούς. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να υπογραμμιστεί αυτό. Πρόκειται για μια σύνοδο κορυφή, το λέω, τον λόμπι των εξοπλισμών. Αυτό κάνουμε, υποτασσόμαστε σε αυτά που περιμένουν από εμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαν να ζούμε σε ένα παράλληλο κόσμο. Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που συγκλονίζεται από την οικονομική κρίση και τι κάνουμε. Συζητούμε για το αν τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε τα κράτη-μέλη στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό ή στον Εθνικό Προπολογισμό μπορούν καλύτερα να αξιοποιηθούν, πιο αποτελεσματικά να αξιοποιηθούν για να αγοράζουμε ακόμη πιο ακριβά, πιο αποτελεσματικά πιο εύχριστα συστήματα όπλων. Και πρέπει να πω ότι δεν εκπλήσουμε ότι τώρα ακριβώς πριν από αυτή τη σύνοδο οι άντες μας λέει δεν μπορούμε να κάνουμε ε, τίποτα, θα απολύσουμε κόσμο γιατί εσείς τα κράτη-μέλη δεν έχετε αναλάβει την δέσμευση που θα, ε, θα έπρεπε για να συνεργαστείτε στην υπόθεση αυτή» και αυτό δεν είναι απλώς ότι ζεύουμε το άλογο προς τα πίσω ή όπως υπόθηκε νωρίτερα, είναι ότι κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι θα πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι τα στοιχεία που αναφέρατε μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε πολύ διαφορετικό τρόπο. Τα 26 δισεκατομμύρια που δίνουμε κάθε χρόνο για τους εξοπλισμούς είναι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο προσφέρουμε ε, για την στήριξη των εθνικών προϋπολογισμών. Θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε έως και 30 δισεκατομμύρια, λέτε. Ναι, ακριβώς αυτό θα οδηγούσε στο να πούν οι πολιτικοί στους εξοπλισμού, εάν μπορούσαν οι πολιτικοί να πούνε στη βιομηχανία εξοπλισμών ότι πρέπει να σταματήσουν πια αυτές τα πάνε. Αλλά το αντίθετο ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή η βιομηχανία εξοπλισμών υπαγορεύει στους πολιτικούς το τι πρέπει να κάνουν. Δεν είστε σε θέση μέσα σε μία δεκαετία να κάνετε τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τη Γερμανία. 30 χρόνια για το Eurofighter. Τι περιμένετε δηλαδή. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς ερχόμαστε εδώ να συμπεριφερόμαστε σαν αθώες περιστερές για να ε, μιλήσουμε για εξοικονόμηση πόρων και πιο αποτελεσματικά συστήματα. Ούτε σε εθνικό, ούτε σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο είναι δυνατόν να καλυφθούν με περισσότερες δαπάνες ή ανάγκες για την άμυνα ή για την προστασία των πληθυσμών. Αυτά είναι τελείως παράδοξα που μας λέτε και θέλω να προειδοποιήσω για, το, για την ασφαλμένη πορεία που έχετε πάρει. Θέλω επίσης να σας ε, επισημάνω το εξής, ότι όσο δεν έχουμε αντιμετωπίσει τις σοβαρές ανισορροπίες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όσο δεν ασκούμε περισσότερη πίεση και κατά τη Ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας ώστε, και αυτή στο βαθμό που συμβάλλει σε αυτές τις ανισορροπίες να αλλάξει συμπεριφορά ώστε να αντιστραφεί αυτή η πλάστιγκα των υπερβολικών εξαγωγικών κερδών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας που είναι εις βάρος των άλλων κρατών δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φάρατζ από το EFT. Well, Ευχαριστώ. Βέβαια είναι Χριστούγεννα τώρα και πάντα μιλάμε για τις 12 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Εγώ θα μιλήσω για τις 21 μέρες και για τα εκατομμύρια ανθρώπων από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Κάτι το οποίο είναι πολύ επίκαιρο στην ε, πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου. Πολύ συχνά εμεί διαμαρτυρόμαστε ότι δεν έχουμε αρκετή επαφή με τον κόσμο. Αυτό όμω θέλουμε να αλλάξει σήμερα. Εδώ ο Βανόρντα από τους συντηρητικούς ήταν ο εισηγητής για την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άνοιξε την πόρτα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να έρχονται και εγώ θα ήθελα να ξέρουν οι Βρετανοί τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς σημαίνει η ελεύθερη κυκλοφορία. Σημαίνει και δωρεάν περίθαλψη, δωρεάν παιδεία, σημαίνει δωρεάν πρόσβαση στα συστήματα ε, πρόνοιας, σημαίνει ελεύθερη πρόσβαση στους εγκληματίες, στις συμμορίες που όλοι τελικά θέλουν να έρθουν στο Λονδίνο που είναι η πιο επιτυχής ε, πόλη στην Ευρώπη η κατάσταση είναι ήδη τόσο άσχημη που 92% των ε, εγκλημάτων που γίνονται στα μηχανήματα που τραβάει κανείς χρήματα ε, προέρχονται από εκεί. Βουλγαρία, Ρουμανία είναι βέβαια άνθρωποι πολύ αξιοπρεπείς οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν ε, καλά αλλά δυστυχώς υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Υπάρχουν συμμορίες από το Βουκουρέστι. Έρχονται στο Λονδίνο, παίρνουν επιδόματα για δύο παιδιά που έχουν και τα χρήματα από τα επιδόματα αυτά είναι πολύ περισσότερα από ό,τι θα έβγαζαν αν στο Βουκουρέστι είχαν μια αξιοπρεπή εργασία. Και γι' αυτό έρχονται στον Ηνωμένο Βασίλειο. Και είναι πολλοί αυτοί. Το έχω πει και συμφωνούν και οι Βρετανοί, φτάνει πια. 80% των Βρετανών δεν θέλουν να αλλάξει κατά σε 21 μέρες και να πάψει να υπάρχει περιορισμό στα σύνορα. Μην ξεχνάμε ότι αυτό θα ενισχύσει την ανεργία των νέων. Και δεν τελειώνει εδώ. Ο Πρωθυπουργός μας, ο κύριος Κάμερον, με την πλήρη στήριξη των εργατικών και των φιλεύθερων, τώρα θέλει η αρχή αυτή των ανοιχτών συνόρων να επεκταθεί, όπως λέει και ο ίδιος, και να πάει από τα... τον Ατλαντικό στα Ουράλια. Καζακστάν, Ουκρανία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα. Το βλέπω. Τόνι Μπλερ τώρα βοηθάει την Αλβανία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, καλή τύχη. Θέλουμε και την Τουρκία να βάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνυμά μας είναι ότι η Τουρκία είναι για χριστουγεννιάτικο δώρο, δεν είναι για την πολιτική ένωση. Δεν θέλουμε ανοιχτά σύνορα. Κύριε Κάμερον, την επόμενη εβδομάδα στη διάσκεψη κορυφής μην παρετηθείτε με τίποτα και προχωρήσετε σε μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Είναι ορολογιακή βόμβα ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Να μην ανοίξουμε την πόρτα και σε έναν ευρωπαϊκό στρατό. Όχι. Θα είναι σεισμός για την ευρωπαϊκή πολιτική. Ευχαριστώ. Ε, κύριε συνάδελφε, ο συνάδελφος Μπρόντς έχει μια ερώτηση. Τη δέχεστε.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 λέστε ε, ή μάλλον υπενήσεστε ότι είστε κατά, είστε κατά της μετανάστευσης. Στις 4 ε, Μαΐου 2010 είπατε ότι ε, εκδίδονται στη Μεγάλη Βρετανία 250.000 άδειες εργασίας. Πριν από λίγο αναφερθήκατε στους Ρουμάνους και τους καταλογίσατε ε, παραβατικές πράξεις στα ATM. Εσείς είπατε, θα μπορούσατε να είσαστε ακόμα πιο συγκεκριμένο. Ρουμάνοι, καταγωγής, Ρουμάνοι, Ρωμά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω κάτι ε, ξεκάθαρο. Το Ενωμένο Βασίλειο δεν είναι κατά της μετανάστευσης. Ε, να καλωσορίσουν. Ε, ε, θέλουμε όμως ένα σύστημα μετανάστευσης ε, που να βασίζεται όπως συμβαίνει στην Αυστραλία σε ανθρώπους με δεξιότητες. Δεν θέλουμε ανθρώπους που έχουν μολυσματικά νοσήματα, δεν θέλουμε άτομα με βεβαρημένο ποινικό μητρό και θέλουμε να μπορούμε να αποφασίζουμε εμεί στο ποιό έρχεται. Εμείς ε, δεν κάνουμε διακρίσεις, ε, δεν δημιουργούμε αποδιοκομπέους τράγου. Απλά και μόνο θέλουμε να ελέγχουμε τα σύνορά μας και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό ω μέλη αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. So. Και τώρα πέθαμε πάλι στη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η κυρία Λεπέρνα Ζητή συγγνώμη δεν μπόρεσε να έρθει. Και τώρα το λόγο έχει ο συνέλφος κύριος Μπρόκ για το ΕΛΚ. Ε, ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Δύο λόγια για την Ουκρανία. Όποιος είδε τι συνέβη σήμερα το βράδυ, και ότι και οι πρωτοβουλίες της κυρίας Άστον των Αμερικανών δεν έφεραν αποτέλεσμα. Νομίζω μπορεί να διαπιστώσει ότι η κατάσταση πάει προς τα χειρότερα. Η πιέση της Ρωσίας, οι πιέσει της Ρωσίας κλέβουν από ένα λαό ολόκληρο τις ελευθερίες του και τα δημοκρατικά του δικαιώματα. Κάτι το απαράδεκτο. Πρέπει να το πούμε αυτό. Συμφωνώ με την κυρία Χάρμς ότι αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δεν έχουμε κοινή πολιτική για τη Ρωσία. Τα ζητήματα που προκύπτουν για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της κοινή Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας είναι πολύ σημαντικά. Γιατί ναι, είμαστε υπέρ του ΝΑΤΟ και πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η διάσταση της ασφάλειας που προσφέρει το ΝΑΤΟ, αλλά πρέπει και να αναπτύξουμε τις δικές μας δυνατότητες, να τις αξιοποιήσουμε για να υπάρχει και ευρωπαϊκή βιομηχανία όπλων και επιλογές ανεξάρτητες από πού θα εξοπλιζόμαστε. Εάν λοιπόν θέλουμε μία συμμαχία των ε, διατεθειμένων να προχωρήσουν, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Αλλά όχι με έναν στρατό γραφειοκρατών που θα περιορίσει κανουμε και αυτο αλλα οχι με εναν στρατογραφιο κρατών που θα περιοριζει δυνατοτητες Με μια κατανομή εργασίας, με μια συνένωση των δυναμιών μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε δηλαδή οι Αμερικανοί να αναλαμβάνουν δράση μέσω του ΝΑΤΟ για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία ή στην ευρωπαϊκή γειτονία. Δεν θέλουμε να γίνει όπως η βρετανική πολιτική, η ευρωπαϊκή, το κανείς, το σκυλάκι της αμερικανικής πολιτικής στα θέματα της άμυνας. Δεν θέλουμε να είμαστε global payer, αλλά global player, όχι να πληρώνουμε, αλλά να καθορίζουμε τα τεκτενόμενα στον κόσμο. Και χρειάζεται γι' αυτό μια κοινοτική πολιτική. Έχουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σταθεί και ταχθεί υπέρ του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, υπέρ του εις 6 μέτρων, Έχουμε κάνει ό,τι χρειαζόταν από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σταθεροποίηση, για τι μεταρρυθμίσει στα κράτη-μέλη και ε, αυτέ τι μεταρρυθμίσει που πρέπει να ενισχυθούν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτό το οποίο ορίζει κατευθυντήριε γραμμέ με τη συναπόφαση και με τι επαφέ του με τα εθνικά κοινοβούλια μπορεί να συναποφασίσει, να συμπροσδιορίσει καλύτερα τα εθνικά προγράμματα που πρέπει να αναπτυχθούν και να αποφασιστούν και το που υπάρχουν εθνικά ζητήματα μπορεί να ενισχύσει την εμπλοκή, το ownership όπως λέμε των εθνικών κοινοβουλίων στα τεκτενόμενα. Αλλά δεν πρέπει να ξεκινήσουμε μια, έναν αγώνα ανταγωνισμών για, για, τα για την κοινωνική προστασία και τα δικαιώματα. Και κάτι ακόμη κύριε Πρόεδρε, δύο λόγια. Με τον κύριο Φαράζ και τα όσα άκουσα. Δεν είναι ούτε ευρώ ούτε μετανάστευση. Απλώς φτηνός λαϊκισμός τίποτε άλλο εις βάρος των ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάθε μέσον να βοηθήσει αυτούς που δεν έχουν ε, θέση εργασίας, αυτούς που μένουν ε, απροστάτευτοι ε, κοινωνικά ή από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη πρέπει να τους προστατέψει. Και είναι καθήκον και της Βρετανίας εφόσον είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το συνεχίσει αυτό. Δεν πρέπει να ακούγονται τέτοιοι λαϊκισμοί. Στο Ευρωπαϊκό ευχαριστούμε. Ο κύριος μου θέλει μια ερώτηση. Δέχεστε μια μπλε κάρτα λοιπόν. Δέχεστε να απαντήσετε. Παρακαλώ. Δέχετε το λόγο. Ευχαριστώ που δέχεστε την ερώτησή μου. Κύριε Μπρόκ, άκουσα ότι είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει ικανότητες πολλές φορές. Τι εννοείτε, εννοείτε ότι θέλετε έναν ευρωπαϊκό στρατό, έναν ευρωπαϊκό στόλο, ευρωπαϊκές αεροπορικές δυνάμεις. Κύριε Μπρόκ, Απαντήστε, παρακαλώ. Αξιότιμη συνάδελφα. Προϋπόθεση νομική δεν υπάρχει, βάση νομική δεν υπάρχει. Αλλά η συνθήκη, η συνθήκη της Λισαβόνας μιλάει για εξασφάλιση κατανομής εργασίας και καλύτερης ε, χρήσης των δυνατοτήτων. Δεν μπορούμε, παραδείγματι, να ε, προχωρήσουμε σε διάθεση ε, γερμανικών στρατευμάτων σε ένα κοινό ευρωπαϊκό ε, εγχείρημα εφόσον υπάρχει εφόσον δεν δίνει την έγκρισή του το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Αλλά με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία μπορούμε να συνδυάσουμε καλύτερα τις δυνάμεις μας. Εσείς μπορεί στο Ηνωμένο Βασίλειο να θεωρείτε ότι μπορείτε να χρηματοδοτείτε ανεξάρτητα την αμυνά σας, αλλά πιστεύουμε εμείς ότι το pooling and sharing όπως το λέμε, η συγκέντρωση δηλαδή πόρων και η κατανομή εργασίας και καθηκόντων είναι η καλύτερη λύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναπτύξουμε και τη δυνατότητα δράσης και να προστατεύσουμε καλύτερα τους λαούς μας κατά τρόπο που μόνιμα δεν θα μπορούσαμε ο καθένας να το πράξει. Είμαστε μικροί ο καθένας χωριστά στο παγκόσμιο σκηνικό. Η Ευρώπη όμως είναι μεγάλη. Ευχαριστούμε. Δύο λεπτά τώρα. Το λόγο έχει ο κύριος Γκουαλιέρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να πω ότι το κοινοβούλιο αυτό το θα επαγρυπνήσει έτσι ώστε οι απόψινές ε, συμφωνίες ε, θα γίνουν απόλυτα σεβαστές. Ε, ύστερα οι συμβασιακές συμφωνίες που φαίνεται να είναι το μοναδικό αποτέλεσμα μιας άσκησης που στόχο είχε να κάνει ένα οδικό χάρτη για την Οικονομική Ένωση. Λίγο μου φαίνεται. Έχουμε την εντύπωση ότι μια πραγματική συμφωνία για τις βασικές αρχές αυτού του μέσου δεν υπάρχει. Μια ενδυναμω, ένας ενδυναμωμένος Επομένω, ε, ε, ε, συντονισμό μπορεί να γίνει μόνο με βάση κίνητρα. Οι χώρε μέλη όμω δεν μπορούν να γνωρίσουν το μηχανισμό αλληλεγγύη. Έτσι, με τη συνήθη στρατηγική των δύο χρόνων, θέλουμε μια συμφωνία για, αυρί, για τι αυρινέ συμβάσει, ενώ τα αποτελέσματα τα δούμε αύριο. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία όμω που έχει μια σύμβαση πολιτικά δεσμευτική, όπω λέγεται, δίχω κίνητρα. Αυτό δεν είναι σαφέ, που δεν είναι. Η όλη συμβασιακή λογική δεν είναι πιστική. Μία λογική διμερούς χαρακτήρα που διατρέχει τον κίνδυνο να είναι ισχυρή με τους αδύναμους, αδύναμη με τους ισχυρούς. Υπάρχει έλλειψη της κοινωνικής διάστασης αυτής της άσκησης. Επιμένουμε επί των πολιτικών προσφοράς όταν η κρίση είναι μια, πολιτι... μια κρίση συζήτηση. Στην ουσία λέμε, λέμε ότι θα, αποφυ... αποφασίσουμε ομόφωνα για θέματα που είναι αποτέλεσμα συναπόφασης. Θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση απόφαση. Εμεί είμαστε έτοιμοι να διαδραματίσουμε το θεσμικό μα ρόλο. Εάν οι αρχέ όμω που αναφέρονται στο ψήφισμα που θα εγκρίνουμε δεν θα, είναι, δεν θα ληφθούν υπόψη, οι συμβασιακέ συμφωνίε, εάν έχουν, ε, πάρουν το πράσινο φω, ε, θα έχουν πολύ δύσκολη ζωή σε αυτό το κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε. Για δύο λεπτά τώρα έχει το λόγο ο κύριος Βότσον. Πρόεδρε, το σώμα πρέπει να εκφράσει την ικανοποίησή του για την δέσμευση για κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας από πλευράς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι κάτι θετικό και ανταποκρίνεται στη δέσμευση του Συμβουλίου. Είναι μια επιτυχία και δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το στρατιωτικό θέμα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι μοιραζόμαστε ένα κοινό στόχο. Μια λοιπόν αποτελεσματική πολιτική έτσι θα συνδυαστεί με την τεχνολογική βάση που διαθέτουμε με χρήματα από τον, ε, το πρόγραμμα Ορίζοντας και έτσι θα έχουμε περισσότερη αναπτυξιακή βοήθεια, δικαιοσύνη, θα υπάρξει νέα ισορροπία μέσα στο ΝΑΤΟ μέσω μιας εταιρική σχέσης εμπορίου και επενδύσεων. Επίσης μια στρατηγική για τη θάλασσα, για τον κυβερνοχώρο και για τα δορυφορικά συστήματα πρέπει να είναι προτεραιότητα για μας. Όσον αφορά τώρα τα μη πανδρομένα σκάφη, για να δούμε σε τι βαθμό ενισχύουν την άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίσης θα πρέπει να ξεχάσει την ενεργειακή πολιτική, να μην είναι μια υποσημείωση. Το να περάσουμε από τα ορεκτά καύσιμα στην καθαρή ενέργεια είναι κάτι ζωτική σημασία για να υπάρχει ασφάλεια, για την προστασία του περιβάλλοντο αλλά και για ανεξαρτησία ενεργειακή από τη Ρωσία. Το Συμβούλιο θα είναι πολύ σοφό αν δεν ακολουθήσει τη συμβουλή του κ. Σβόμποντα. Ο κ. Σβόμποντα τα έβαλε με την πολιτική του Όλη Ρεν που θέλει να βάλει μια ισορροπία στα λογιστικά τη Ευρώπη. Βλέπουμε όμως τι βάρος επομίζονται τα κράτη-μέλη. Τι θέλει, να καταδικάσουμε τα παιδιά μας να πληρώνουν τα χρέη των γονιών τους, να εφαρμόσουμε του Μπόρντον Μπράουν και του Σαπατέρου και του Ολάντα τις πολιτικές. Κύριε Σφόποντα, σε αυτή την περίπτωση οι φιλελεύθεροι θα δείξουν τι εξίζουν στην προεκλογική εκστρατεία εν ώψη των ευρωεκλογών. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Βότσον. Δύο λεπτά τώρα το λόγο έχει η κυρία Κρόνμπεργκ. Αξιότιμα μέλη, οι δαπάνε για την άμυνα περιορίζονται και αυτό επηρεάζει άμεσα τι αμυντικέ μα ικανότητε. Παρόλα αυτά, αυτή η αρνητική πτυχή μα πλήττει ακόμα περισσότερο λόγω του περιορισμένου συντονισμού και συνεργασία μεταξύ ημών των Ευρωπαίων. Η ομάδα μα πιστεύει ότι η ασφάλειά μα, η εθνική, εξαρτάται από την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Συνεπώ, θα επιθυμούσαμε να ζητήσουμε από τι χώρε μέλη να στηρίξουν τι ευρωπαϊκέ ευρωπαϊκές αμυντικές ικανότητες, να αποφευθούν οι επικαλύψεις. Του ζητάμε να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικές οι βιομηχανίες για να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός. Χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό εξάμεινο για θέματα ε, ε, ασφάλειας και άμυνας. Θα πρέπει να υπάρξει εναμόρυση των προτύπων και της πιστοποίησης των μηχανισμών ασφάλειας, των εξοπλισμών ασφάλειας. Αυτό που δεν θέλουμε είναι εξαγωγή όπλων που να γίνεται αυτόματα ε, ε, ε, όπλα που είναι κανένα να σκοτώσουν χωρίς την εμπλοκή των ανθρώπων. Θα πρέπει να υπάρξει ένα καθεστώς ελέγχου των όπλων και θέλουμε να υπάρξει μια γενική συμφωνία αξιότιμη μέλη στο επόμενο συμβούλιο Θέλουμε να ενισχυθεί το αμυντικό πακέτο όπω προτάθηκε στον ανακοινωθέν τη Επιτροπή. Οι χώρε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εντείνουν τη συνεργασία τους και το συντονισμό τους ό,τι αφορά τις πτυχέ αυτέ τη Άμυνα που θα οδηγήσουν σε μια πραγματική πολιτική. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά. Van που πριν από λίγο ανακαλύψαμε ότι είναι ταξιάρχης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την επόμενη εβδομάδα θα συζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να αναλάβει ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός ε, για την ευρωπαϊκή πολιτική Άμυνα. Ακούσαμε ήδη τα μάντρα και τις εποδούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπω ότι το πλαίσιο όμως για την άμυνα, για την προσεχή εβδομάδα, πέραν ενός καταλόγου για τα μαθήματα που έχει να ετοιμάσει στο σπίτι η Επιτροπή, ε, δεν έχει μεγάλο εύρος, ούτε οράματα, ούτε προτάσεις σε σχέση με τα όσα έχουν προταθεί στις 25 Νοεμβρίου. Ερωτώ λοιπόν προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή τι σημαντικές αποφάσεις για την άμυνα πρόκειται να ληφθούν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στο Συμβούλιο την προσεχή εβδομάδα. Διότι εγώ πιστεύω ότι για την κοινή πολιτική, πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας. Έχει πια έρθει η ώρα, διότι και στις ε, πρωτεύουσε των κρατών μελών, αν και κάποιοι ίσως ζουν ε, στο φανταστικό κόσμο της Αλίκης, σε αυτό το κοινοβούλιο, ε, στις χώρες μέλη λοιπόν και τις κυβερνήσεις τους δεν διαγνώσκω καμία βούληση για πρόοδο προς μια ευρωπαϊκή πολιτική και βιομηχανία άμυνας και ασφάλειας, μάλλον προς και πολύ σωστά πολιτικές δράσεις για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ανθρωπιστική δράση. Πολλοί τα ήμασταν που χρόνια τώρα αγωνιζόμαστε για αυτή τη μεταστροφή ώστε να κάνει επιτέλους κάτι χρήσιμο η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπληρωματικά δηλαδή και όχι κατά απομίμηση του στρατιωτικού σκέλους του ΝΑΤΟ. Ε, χρειάστηκε να κάνει αυτό το άλμα η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι έτσι θα θέσει ένα θεσμικό ίχνος ως προς τις δραστηριότητες της άμυνας που όμως δεν θα πρέπει να επικαλύπτονται με τα όσα ήδη κάνει το ΝΑΤΟ. Μελλοντικέ δράσεις της ε, κοινή πολιτικής ασφαλείας και άμυνας θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ήταν κυρίως μη στρατιωτικές, πολιτικής προστασίας δηλαδή. Εδώ είναι σαν να λέμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε τον υδραυλικό χωρίς όμως να υπάρχει νερό. Ευχαριστούμε κύριε Βανόρντεν. Για ένα λεπτό ο κύριος Κουντής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αναφερόμαστε στην επόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού συμβουλίου σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκοί λαοί υποφέρουν από τις πολιτικές λιτότητας της ευρωπαϊκής ένωσης σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές δημοκρατικές και κοινωνικές κατακτήσεις καταργούνται στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και των κερδών. κύριε πρόεδρε στο επόμενο συμβούλιο οι ηγέτες θα μιλήσουν για την οικονομική κατάσταση της ένωσης για την οικονομική κατάσταση της ονε. θα ακούσουμε πάλι πήραμε μια γεύση για την τραπεζική ένωση για το ευρωπαϊκό εξάμεινο για την οικονομική διακυβέρνηση δεν θα ακούσουμε όμως γιατί θα αγνοήσουν για άλλη μια φορά τα αποτελέσματα τα καταστροφικά αυτών των πολιτικών. δεν θα ακούσουμε παραδείγματο χάρη για το 1,5 εκατομμύριο ανέργων στην ελλάδα δεν θα ακούσουμε ότι χιλιάδε νοικοκυριά σήμερα στην ελλάδα δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα ακούσουμε ότι η ελλάδα μια χώρα που βρίσκεται κάτω από τη στενή εποπτεία όλων των θεσμών τη ευρωπαϊκή ένωση οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι και θα συνεχίσουν του εκβιασμού για του πληστηριασμού και τι καταθέσει των ελληνικών νοικοκυριών. κύριε πρόεδρε μια τέτοια ευρωπαϊκή ένωση ένα τέτοιο συμβούλιο τέτοιοι ηγέτε είναι αναντίστοιχοι των εξελίξεων δεν ανταποκρίνονται στα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών. εμεί ω αριστερά θα αγωνιστούμε για ριζικές αλλαγές και ανατροπές για να μπορούμε να μιλάμε για μια ευρώπη της εργασίας της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. ευχαριστώ πολύ. Ενάμιση λεπτό τώρα ο συνάδελφος Πάξας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Συμβούλιο έχει μια ημερήσια διάταξη με πολύ σημαντικά θέματα σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Και θα συζητήσει την ε, ε, Ένωση, την Αμυντική Ένωση και τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί το θέμα Ουκρανίας η Ένωση. Μέχρι στιγμής όμως συγκεκριμένες απαντήσεις δεν έχουν δοθεί. Πρέπει λοιπόν ε, να διαπιστώσουμε ότι δεν έχει γίνει κανένα ανοιξικέλευτο βήμα, τουλάχιστον για φέτος. Ε, δεν έχουν υποστηριχθεί τα μέτρα λιτότητας με, από τις απαραίτητες ε, ε, οικονομικές μεταρρυθμί... τις απαραίτητες οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Μόνο εποχιακή απασχόληση μπορούμε να πούμε, μπορεί να διαπιστωθεί ότι έχει μετριάσει το φαινόμενο της καλπάζουσας ανεργίας. Τα μέτρα ήταν εν γέννη μόνο προσωρινά και τώρα με το χειμώνα που πέφτει και το κρύο τα προβλήματα οξύνονται σημαντικά και θα δούμε πιστεύω τα αποτελέσματα των όσων συμβαίνουν τώρα το καλοκαίρι του χρόνου όταν ε, θα είναι ξεκάθαρη η εικόνα. Πρέπει λοιπόν ιδιαίτερα να αναφερθούμε στα ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις που θα πρέπει να ενισχυθούν, αλλά ταυτόχρονα με τον όρο να απασχολούν ανθρώπους έως 30 ετών. Πρέπει να προσφερθεί ε, ε, ε, υποστήριξη οικονομική στους νέους που για πρώτη φορά ξεκινούν μια πορεία στον εργασιακό βίο ή προσπαθούν τουλάχιστον. Πρέπει να μειωθεί η επιβάρυνση, η φορολογική, στους μισθωτούς. Οι μισθωτές οικογένειες δεν πρέπει να φορολογούνται τόσο πολύ, αλλά το ελάχιστο. Ευχαριστούμε για 1,5 λεπτό τώρα. Κυρία Σίνκλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ συζητάμε για την Οικονομική Ένωση ολόκληρη την Ευρώπη και τι θα αποφασίσει να βάλει στην ημερήσια διάταξη το Συμβούλιο Άμυνα. Εγώ θα έλεγα ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι αυτό είναι ένα από τα τελευταία πράγματα που απασχολεί τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι θέλουν να ασχοληθούμε με την απασχόληση, με το κόστος ζωής τους, ε, με τον πληθωρισμό. Αλλά εσεί δεν θέλετε να μιλήσετε για αυτά. Θέλετε να μιλήσετε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα. Εδώ άκουσα να μιλάτε για τον ανταγωνισμό με τι ΗΠΑ. Μα γιατί είμαστε 28 κυρίαρχα έθνη. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο, καμία ε, πρόθεση να αλλάξει αυτό πρέπει να έχετε τη συνένεση των ανθρώπων. Εσείς όμως δεν θέλετε αυτό, θέλετε να προχωρήσετε και να περάσετε σε αυτό το καθεστώς του σούπερ κράτους. Μα γιατί, γιατί θέλουμε να ε, ξαναφεύρουμε τον τροχό. Έχουμε τον ΝΑΤΟ, υπάρχει, το οποίο έχει αποδείξει την αξία του. Αυτό χρειαζόμαστε, τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα θέλουμε την απασχόληση. Εσείς ε, χαίρεστε που τώρα έχουμε και την ε, Λετωνία στο ενίο νόμισμα. Ναι. Αλλά δεν φτάνει που υπάρχουν τόσα προβλήματα, βάζετε και την Λετωνία. Και τελικά τι θα κάνετε, θα είναι χειρότερα ακόμα τα πράγματα από ό,τι ήταν πριν με το ευρώ. Θα είναι μια χειρότερη ύφεση που θα πονέσει και πάλι τους λαούς της Ευρώπης. Σταματήστε πια. σε ευχαριστούμε. Δύο λεπτά. Ο κύριος Σαουντάργας τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, στις 19 και 20 Δεκεμβρίου θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πώς θα καθοδηγήσει τη μελλοντική πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Θα συζητήσει προτάσεις για πιο αποτελεσματική ΩΝΕ, για ενίσχυση του συντονισμού της οικονομικής, των οικονομικών πολιτικών για να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα οικονομική σταθερότητα. Οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης θα καταγράψουν την πρόοδο και την εφαρμογή των μέτρων για την προαγωγή της ανάπτυξης και της επασχόλησης. Αυτά είναι ασφαλώς τα θέματα που ανταποκρίνονται στις ε, προσδοκίες των Ευρωπαίων. Θα συστήσουν την διαχείριση της Τραπεζικής Ένωσης, επίσης αρχική κρατών και κυβερνήσεων. Αυτό είναι μεγάλη ευθύνη για τη Λεθονική Κυβέρνηση, για τη Λεθονική Κυβέρνηση και την Προεδρία στο Συμβούλιο την ε, θέσπιση ενό ενιαίου εποπτικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση τη ε, κρίση. Ελπίζω δε ότι θα μπορέσει να συμφωνήσει για τι γενικέ ε, διατάξει για το δεύτερο πυλώνα, τον μηχανισμό επίλυση διαφορών, που θα βοηθήσει την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητα των τραπεζών. Δηλαδή θα μπορούν μέσα από το μηχανισμό αυτό οι τράπεζε όταν βρίσκονται σε δυσκολία μόνε του συνεργαζόμενε να λύνουν τα προβλήματά του και έτσι θα είναι ε, θα απαλλαγούν οι πολίτες από αυτό το άχθος ε, και θα αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη στην, ε, στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο. Κύριε Πρόεδρε, επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καταγράψει την πρόοδο σε επίπεδο στον τομέα της ενέργειας έχουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος προβλέπει γραμμή ειδική, κονδύλιο ειδικό για στρατηγικά ενεργειακά έργα και ξέρουμε ότι υπάρχουν τέτοιου είδους έργα που έχει ετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρουσιάζουν ενδιαφέρον ε, κοινό γιατί οι Ευρωπαίοι πληρώνουν πολύ ακριβά την ενέργεια. Πρέπει λοιπόν να μεριμνήσουμε ώστε τα σχέδια αυτά, τα έργα αυτά να υλοποιηθούν σωστά και εγκαίρως για να μειωθούν οι μεγάλες αποκλήσεις τιμές και να μειωθεί βέβαια το κόστος για να έχουμε καλύτερη ανταγωνιστικότητα και βέβαια τα τιμές πιο οικονομικές για τον καταναλωτή. Ευχαριστούμε για 1,5 λεπτό ο κύριος Γκερέρο Σαλόμ τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην αρχή ο κύριος Σβόποντα ηρωνεύτηκε κάπως τα στοιχεία, τα συγκριτικά που έχουμε ανάμεσα στις Ηνωμένε Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απασχόληση. Και είναι θλιβερή η ηρωνία αυτή, γιατί εκεί είναι θετικά τα αποτελέσματα, ενώ εδώ είναι ραχητικά, αρνητικά. Στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάνω από 10 χώρες με απασχόληση, με ανεργία μάλλον τόσο υψηλή που θα χρειαστούν δεκαετίες για να κατέβει η ανεργία στο 10%. Το 2008-2012 και του χρόνου είχαμε πολιτικές πιο αποτελεσματικές στην άλλη πυροπότη στην Ευρώπη. Αυτό δείχνει ότι η λιτότητα δεν έδωσε τα θετικά αποτελέσματα που δίνουν άλλες πολιτικές που χρησιμοποιούνται σε άλλους χώρους. Και δεν πρόκειται εδώ πέρα μόνο για τις διάφορες πολιτικές, πρόκειται και για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Λαμβάνονται οι αποφάσεις εδώ τη μία μέρα για την επόμενη όταν καταφέρουμε να έχουμε μια γρήγορη πολιτική συμφωνία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι αλήθεια ότι είχαν και αυτές το shutdown, δηλαδή παράλυσε το κράτος για κάποιους μήνες εκεί. Όμως, ας έρθουμε πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα ακόμα συζητάμε τον μηχανισμό τραπεζικής εξυγένσης και δεν γνωρίζουμε κατά πόσο θα επιτευχθεί ή όχι συμφωνία στο επόμενο Συμβούλιο. Όμως τα δεδομένα δείχνουν ότι το ενίο Ταμείο Εξυγένσης θα χρειαστεί 10 χρόνια ή το 2026. Με ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να έχουμε μια πραγματική τραπεζική ένωση που να βοηθήσει στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομίας. Άρα χρειάζεται να αλλάξουμε πολιτικές. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις για τις πολιτικές αυτές στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε Ενρίκε. Για δύο λεπτά ο κύριος Νταφ τώρα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρόκειται να συμφωνήσει επί ενός εκτενούς καταλόγου θεμάτων που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει και θα έπρεπε να κάνει είναι να υιοθετήσει μια απόφαση σε ό,τι αφορά την Κεντρική Αφρική για να υποστηρίξει τα γαλλικά στρατεύματα. Εγώ επισκέφθηκα την περιοχή και θα πρέπει να πω ότι αποτελούν ένα εξαιρετικό παράδειγμα στρατιωτικής συνεργασίας. Στο παρελθόν από το 2005 δεν είχε υπάρξει ανάπτυξη αυτών των στρατευμάτων, από τότε δηλαδή που δημιουργήθηκαν. Λόγω της άσκησης ε, του ΒΕΤΟ πρώτα από πλευράς της Γερμανίας και μετά από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου. Την ερχόμενη εβδομάδα μας δίνεται η ευκαιρία να υπάρξει να υπάρξουν μέτρα έτσι ώστε θα αρχίσουμε να υιοθετούμε συλλογικές δράσεις οι οποίες θα οδηγήσουν στην προώθηση των συμφερόντων στον τομέα της ασφαλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Άντριου. Η κυρία Τζιλ Εύανς τώρα για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν θέλουμε η Ευρώπη να είναι λειτουργική, θα πρέπει να δείξουμε ότι μπορεί να διαδραματίσει στο μέλλον ένα διεθνή ρόλο θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε στην ειρήνη. Μια πραγματική πολιτική ασφάλεια θα πρέπει να συνοδεύσει τις πολιτικές για φτώχεια, ε, για την ενέργεια κτλ. Θα πρέπει πρέπει να κινηθούμε προς τον τομέα της κατάκτησης της ειρήνης. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με τον πολιτικό και όχι με το στρατηγικό σκέλος. Θα πρέπει να προωθήσουμε την κατανόηση και να προλάβουμε τις συγκρούσεις σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Ήρθε η ώρα για να επενδύσουμε όχι στα όπλα αλλά στους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους για να βρουν μια θέση εργασίας, για να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι όλοι οι λαοί της Ευρώπης όλες οι χώρες να διαδραματίσουν ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου. Ευχαριστούμε κύριε Εύανς. Τώρα ο συνάδελφος Τοσονόφσκι για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου θα είναι η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης, η οποία απασχολεί περί τα 400.000 εργαζομένους. αλλά οι κίνδυνοι σχετικοί με την ασφάλεια αλλάζουν διαρκώς στον κόσμο. Είναι πιο πολλές οι ανθρωπιστικέ παρεμβάσει. Είναι πιο μεγάλη η κίνδυνη της δημοκρατία. Όλα αυτά σημαίνουν νέες προκλήσεις και σε τεχνικό επίπεδο. Πολλά κράτη-μέλη πρέπει να λάβουν, να λάβουν μέρος στη φάση της προετοιμασίας και της ανάπτυξης. Και χρειάζεται η μέγιστη δυνατή τεχνολογική συμβατότητα, η βέλτιστη χρήση των πόρων, των κοινών πόρων και σε μια εποχή οικονομικής λιτότητας και λιτότητας, μείωση κόστους λειτουργίας ή επιχειρησιακού. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μειώσει τις εξαρτήσεις της από χώρες ξένες και θα ενισχυθεί το δυναμικό για την άμυνά μας στο μέλλον. Επιμένω λοιπόν ότι χρειάζεται μέγιστο συντονισμό των υφισταμένων μέσων με τον ΝΑΤΟ. Ευχαριστούμε συνάδελφε. Η κυρία Μαρίσα Ματίας τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πρόεδρε, οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου είναι όλο και περισσότερο συναντήσεις μεταξύ λόμπι. Ή, εν πάση περιπτώσει, τα λόμπι καταφέρνουν και εισβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο ανταποκρίνεται όλο και λιγότερο στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Χρόνο με το χρόνο εξετάζουμε τα οικονομικά ζητήματα και το Δεκέμβριο αποφασίσαμε να δώσουμε το λόγο στα λόμπι της άμυνας, των εξοπλισμών. Ενώ οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν άλλα προβλήματα. Λέμε πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα στον αμυντικό εξοπλισμό και την αμυντική πολιτική. Μα δεν είναι αυτό το πραγματικό πρόβλημα των πολιτών οι οποίοι ζουν υπό συνεχή λιτότητα, με ένδια, με προβλήματα υγείας εκπαίδευσης και έπειτα, Πρόεδρε. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς μπαίνει σε ένα δρόμο χωρίς επιστροφή. Θυμάμαι έτσι μια ταινία του James Bond, όπου έλεγε ότι θα το καταστραφεί το εγχείρημα σε λίγο μόνο χρόνο. Ευχαριστώ κύριε Σαλαβράκο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε βέβαια κάπως σταθεροποιείται η οικονομική κατάσταση στην ευρώπη και συμφωνώ σε αυτό αλλά ανάπτυξη δεν βλέπουμε. οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες κλείνουν η μια μετά την άλλη και επενδύσεις δεν γίνονται στην ευρώπη. το ερώτημα είναι υπάρχουν στοχευμένες δράσεις στην επιτροπή και το συμβούλιο για αντιμετώπιση του προβλήματος. μιλήσαμε για την ουκρανία. οι πολίτες εκεί αναζητούν την ευρωπαϊκή ένωση. στην ευρώπη αυξάνεται ο ευρωσκεπτικισμός μας προβληματίζει. μιλάμε σήμερα για κοινή πολιτική άμυνα στην ευρώπη και πολιτικές απασχόλησης. την ίδια ώρα η τρόικα στην ελλάδα επιμένει στο κλείσιμο των πολεμικών βιομηχανιών και την απελευθέρωση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας γεγονός το οποίο δεν έχει κανένα άμεσο ουσιαστικό οικονομικό αποτέλεσμα. μόνον επιδότηση του ευρωσκεπτικισμού κάνει ερώτημα προτίθεστε να παρέμβετε στην τρόικα ώστε να αποσυρθούν οι περίεργες αυτές αξιώσεις τους για την ελλάδα; ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Επίσης για ένα λεπτό τώρα έχει το λόγο η κυρία Στάσεν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζει Σκέφτεται μάλλον ότι πρέπει κάτι να αλλάξει και σκέφτεται ότι πρέπει να αλλάξει το θέμα της άμυνας. Οπότε γίνονται σχέδια για στρατεύματα ευρωπαϊκά που θα αναπτυχθούν και θα προχωρήσουν σε, κοινές, ε, σε κοινά χειρήματα. Όμως όλα αυτά πληρώνονται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Από τα χρήματα του φορολογούμενου που πετιώνται τελικά για να ενισχυθεί η γραφειοκρατία θέλει να γίνει υπερδύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτες όμως δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτά τα χόμπι. Διότι από πίσω τι κρύβεται, κρύβεται η δημιουργία ενός ομοσπονδιακού κράτους. Πρόεδρε, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε αλλιώ. Πρέπει να φροντίσουμε τα θέματα αυτά να γίνονται είτε διμερό είτε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και όχι σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω λοιπόν η διάσκεψη κορυφή να το καταλάβει αυτό και να μην προχωρήσει. Αλλιώ θα είναι μεγάλη απογοήτευση και δεν θα είναι προ το συμφέρον τη Ολλανδία. Και κύριε Μπρόκο, μιλάτε για λαϊκισμό. Μα η μεγάλη κρίσιμη καμπή για την Ευρώπη θα είναι οι επόμενες ευρωεκλογέ. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σε ευχαριστούμε. Για δύο λεπτά τώρα το λόγο έχει ο κύριος Λαβία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, κύριε Υπουργέ, το επόμενο Συμβούλιο θα αποτελέσει μια ευκαιρία για τους επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων ε, να κάνουν ε, ορισμένες σκέψεις εν ώψη των αποφάσεων που θα πρέπει να λάβουν τους επόμενους μήνες για να αυξήσουν τις προσπάθειες ε, προς την κατεύθυνση της ανάκαμψης ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χώρες μέλη που, που καταβάλουν προσπάθειες εξυγίανσης δεν θα πρέπει να μας κάνουν να ξεχνάμε ότι η έξοδος από την κρίση είναι η ανάπτυξη και όχι ε, η λιτότητα. Μια ανάπτυξη που βασίζεται σε στοχευμένους τομείς. Δεν είναι εποχή για λιτότητα, είναι εποχή για να αλλάξει η πορεία μας προς μια νέα πολιτική που θα είναι σε θέση να δώσει όθηση στην οικονομία. Θα πρέπει να ανανεωθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις εξουσίες της Federal Reserve θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στις χώρες μέλη να επενδύσουν στην ανάπτυξη για να μπορέσουν να ε, προφυλάξουν τους σπόρους τους στον τομέα της πολιτικής άμυνας. Πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή να αφήσουμε ε, τις, ε, τους, προσωρινούς, τους προσωπικούς εγωισμούς και να χρησιμοποιήσουμε τις ικανότητες της κάθε χώρας μέλους, δαπανώντας λιγότερο, δαπανώντας όμως με έναν τρόπο περισσότερο αποτελεσματικό και καταρτίζοντας έναν οδικό χάρτη με συγκεκριμένες προθεσμίες για να υπάρξει ένας ε, να υπάρξουν συντονισμένες κινήσεις στον τομέα της άμυνας. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, πρωτοβουλία που ελήφθη μετά τα τραγικά συμβάντα στη Λαμπεντούσα. Η πρωτοβουλία αφορούσε τις ε, τον έλεγχο των περιπολιών. Χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία το θέμα της μετανάστευσης δεν θα, φορεί, θεωρείται ένα μεμονωμένο φαινόμενο αλλά ένα διαρθωτικό φαινόμενο που αφορά τη σμήλη εισόδου όλη της Ευρώπης. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι προειδοποίηση για όλους. Αυτοί που είναι έξω θέλουν να μπουν ενώ εμείς που είμαστε μέσα δεν έχουμε αποφασίσει να αλλάξουμε πορεία για μια διαφορετική Ευρώπη για να υπάρχει περισσότερη Ευρώπη που θα μας βοηθήσει να βγούμε από την κρίση. Ευχαριστούμε κύριε Λαδία, Η κυρία Κοπάχη. τώρα για δύο λεπτά. Έχουν περάσει δέκα χρόνια από το 2003 όταν αποφασίστηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας και πέντε χρόνια από τη συζήτηση για την εφαρμογή της. Για το λόγο αυτό η συζήτηση για την άμυνα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου είχε καλλιεργήσει πολλές φιλοδοξίες. Με μεγάλη πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στείλαμε στην προηγούμενη Ολομέλεια ένα ισχυρό μήνυμα ότι πρέπει να προχωρήσουμε και στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας ότι η κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας είναι συστατικό στοιχείο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ότι αν δεν προχωρήσουμε η ένωση δεν θα μπορέσει να διαδραματίσει το ρόλο της ως διεθνής δρόμου και πάροχος ασφάλειας και θα παραμείνει μόνο μια μεγάλη αγορά. τονίσαμε ότι η οικονομική κρίση οδήγησε σε αναγκαίες περικοπές και στον αμυντικό προπολογισμό των κρατών μελών υποχρεώνοντάς μας να κάνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους και ότι η λύση είναι συντονισμός συνεργασία και οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων. είπαμε ότι η κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας πρέπει να γίνει ορατή ότι δεν μπορεί να είναι αντικείμενο συζήτησης σε επίπεδο ελίτ αλλά ότι χρειάζεται τη συμμετοχή και στήριξη των πολιτών. προτείναμε συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογή των προβλέψεων της συνθήκης της λισαβόνας για μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία για το start up fund ή το άρθρο 44 για εντολή σε ομάδα κρατών μελών να λαμβάνουν συγκεκριμένες αποστολές. Ζητήσαμε τη θεσμοθέτηση Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας, τακτικές συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οδικό χάρτη για τα επόμενα βήματα. Δυστυχώς, από ό,τι έχουμε δει ως τώρα, τίποτα από όλα αυτά δεν θα συμβεί πέρα από την υιοθέτηση των πέντε πιλωτικών προγραμμάτων πέρα από την υπόσχεση για επανεκτίμηση της κατάστασης τον ιούνιο του δύο τίποτα συγκεκριμένο γενικόλογες αναφορές και αναμάσιμα γνωστών συνθημάτων για τη σημασία της άμυνας. η έλλειψη πολιτικής βούλησης η ατολμία οι εθνικοί εγωισμοί φαίνεται ότι επικρατούν για άλλη μια φορά και οδηγούν το ευρωπαϊκό συμβούλιο στον κατώτερο δυνατό παρανομαστή. είναι κρίμα και εδώ η λύση είναι περισσότερη και όχι λιγότερη ευρώπη αλλά τα κράτη μέλη δειλά αναβάλουν για το μέλλον αναγκαίες αποφάσεις μεγάλες αποφάσεις. επαναλαμβάνω είναι κρίμα. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Για δύο λεπτά τώρα έχει το λόγο ο κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να είμαι πολύ ξεκάθαρος απέχουμε έτη φωτός από έναν Ευρωπαϊκό στρατό. Η δική μου γενιά τουλάχιστον δεν πρόκειται να ζήσει την ε, δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού στρατού. Για να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα θα πρέπει πολλά και διαφορετικά προσκόμματα να αντιμετωπιστούν. Πρόκειται για πολιτικά, για οικονομικά αλλά και για τεχνολογικού χαρακτήρα προσκόμματα. Είναι μια πηγή ε, σύγχυσης όμως και απαράδεκτης ε, σπατάλης ο κατακαιρματισμός της ε, αμυντικής βιομηχανίας και δράσης. Αυτό σημαίνει και μεγαλύτερο κόστος και χειροτερό συνδυασμό των πόρων για την έρευνα και την καινοτομία. Δηλαδή δεν έχουμε την οικονομία κλίμακας. Είναι ένα πρόβλημα γνωστό, ανέκαθεν, και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Για τους λόγους που ανέφερα τώρα ο Ευρωπαϊκός στρατός, ε, μια βιομηχανία δηλαδή αποδιαρθρωμένη, πρέπει να αρχίσει τουλάχιστον να διαφαίνεται στον ορίζοντα. Τον ορίζοντα αυτόν ο Ντεγκόλ τον είχε περιγράψει με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Μας έλεγε ότι ο ορίζοντας όσο προχωράμε τόσο υποχωρεί. Άρα λοιπόν τι θα κάνουμε, θα περιοριστούμε σε πιο μετριοπαθείς στόχους λίγα μόνο κράτη-μέλη με τον κατάλογο, μέσα στον κατάλογο των ε, δυνατοτήτων, περισσότερα κράτη-μέλη στην εξάσκηση και στο προσωπικό. Ίσως αυτό δεν είναι μια κακή λύση για να αναπτυχθεί η διαλειτουργικότητα των δυναμιών μας, των δυναμιών κρούσεως. Αλλά το πρόβλημα είναι πάνω απ' όλα πολιτικό. Δεν έχει κανένα νόημα να δείχνουμε ως πρόβλημα την ανεπάρκεια του δυναμικού όταν τα κράτη-μέλη διχάζονται αμέσω μόλις ε, ζήτημα παρέμβασης όπως στο Μαλί επί παραδείγματι όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να επιδείξει ή να αποδείξει ότι δεν έκανε διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει μέσα που έχει στη Ευχαριστούμε Σάρλο. Για ένα λεπτό τώρα έχει το λόγο ο κύριος Eichhout. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε ότι η άμυνα θα είναι το κεντρικό σημείο στην επόμενη διάσκεψη κορυφής. Θα μιλήσουν οι ηγέτες κατών και κυβερνήσεων για την αμυντική βιομηχανία. Υπάρχει βέβαια και το οικονομικό ζήτημα και αυτό θα είναι στην ημερήσια διάταξη. Έχουν τεθεί βήματα, όπως και χτες έγινε με το ΕΚΟΦΗΝ, έτσι και τώρα, για ένα ταμείο εξυγίανσης, το οποίο όμως οργανώνεται διακυβερνητικά. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα είναι στην ημερήσια διάταξη οι διμερείς συμβάσεις ανάμεσα στις χώρες μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. τυφλή, λοιπόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το Δημοκρατικό Έλεγχο που πρέπει να υπάρχει πάνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία παίρνει όλο και περισσότερη εξουσία κάνει και περισ... όλο και περισσότερο έλεγχο. Πότε επιτέλους θα καταλάβουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ελέγχεται δημοκρατικά. Τέλος, όσον αφορά την κοινωνική Ευρώπη, εδώ υπάρχουν δύο αδύναμες παράγραφοι για αυτήν. Πότε λοιπόν οι ηγέτες κατών και κυβερνήσεων θα καταλάβουν ότι το μέλλον της Ευρώπης θα είναι κοινωνικό ή δεν θα υπάρχει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Για ένα λεπτό τώρα έχει το λόγο η κυρία Άντερσον. Κύριε Πρόεδρε, το μίλημά μου προς ε, τους ε, πολίτες ε, που βρίσκονται στο μνημόνιο στην Ιρλανδία είναι το εξής. Μην πιστεύετε να σας πούνε ότι είναι επιτυχημένο το μνημόνιο, γιατί είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση όπου τα ψέματα καλύπτουν την αλήθεια. Η αυξανόμενη ανεργία, η αναγκαστική μετανάστευση είναι η αποδιάρθρωση κοινωνική είναι τα κατάλοιπα της Τρόικα, είναι η κληρονομιά της Τρόικα με την κυβέρνηση η οποία με πολύ μεγάλη χαρά ακολουθεί τις περικοπές και την πολιτική λιτότητα που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταστροφικά λοιπόν τα αποτελέσματα για την οικονομία της Τρόικας αλλά και άλλων κρατών που βρισκόνται στο μνημόνιο, της Ιρλανδίας αλλά και άλλων κρατών που βρισκόνται στο μνημόνιο με τις επιταγές της Τρόικα αντί να αναλάβουμε μέτρα με πιο φιλόδοξο ε, πλαίσιο, με πιο φιλόδοξο ορίζοντα ε, παρά τις φωνές που ακούγονται εδώ στο Κοινοβούλιο για περισσότερη και πιο καλή ε, ρύθμιση των προβλημάτων. Είναι ε, τρομακτικό το να λέει ότι πρέπει να γίνουν και άλλες περικοπές και άλλες ε, οικονομίες. Ενώ ταυτόχρονα προχωρούμε προς την περισσότερη στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εξοπλισμούς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χαντς Πέτερ Μάρτιν τώρα έχει το λόγο. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Θα προσπαθήσω να μιλήσω πολύ σιγανά, εάν μπορείτε να με ακούσετε. Δεν είναι ανοησία το να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια πορεία προεκλογική. Ούτε είναι λάθος το να πούμε ότι κινδυνεύουμε το προσεχές κοινοβούλιο να ε, έχει στους κόλπους του μια ισχυρή ακροδεξία ομάδα. Εδώ λοιπόν αυτό πρέπει να σημάνει κόδωνα κινδύνου σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να διαρωτηθούμε τώρα είναι η στιγμή να μιλήσουμε για την άμυνα, να προβάλλουμε την κοινή άμυνα και να ξεχάσουμε τα κοινωνικά θέματα. Είσαστε τελείως, τελεία, τελεία, τελεία, ερωτά ο πολίτης της Ευρώπης. Ο πολίτης της Ευρώπης ο οποίος βλέπει το Συμβούλιο, την Επιτροπή, εσάς εδώ τους συναδέλφους να δαπαρώτε τόσα λεφτά και αισθάνετε τόση ανησυχία και λέει «Μα αυτοί μπιπ μπιπ μπιπ κάνουνε, είναι δυνατόν εσείς να συνεχίζετε, μα δεν είναι αγάπια, κάντε κάτι». Για δύο λεπτά τώρα. Ο Ζων Πιέρ Οντί, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι πρώτες μου λέξεις είναι για να εκφράσω τη λύπη μου για την απρουσία του Προέδρου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πραγματικά δεν ξέρω, δεν τον καλέσαμε ή αρνήθηκε να έρθει. Δεν έχουμε πλέον σχέση με τους επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων. Συναντάτε το Συμβούλιο. Εγώ δεν αμφισβητώ τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Γενικών Υποθέσεων. Απλά και μόνο εκφράζω τη λύπη μου για την απουσία του Προέδρου. Σε αφορά την ε, ευρωπαϊκή πολιτική άμυνα, είναι ένα τομέα με ιδιαίτερη ζώντα χαρακτηριστικά που έχει υποχρεώσει σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα συστήματα και ε, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική άμυνα, βιομηχανία τη άμυνα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την ανακοίνωσή τη. Ε, Εμεί προτείναμε την ε, δημιουργία ενός οικονομικού φορέα για να έχουμε την βεβαιότητα σε ό,τι αφορά την απασχόληση, σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση της παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και για να μπορέσουν να υπάρξουν κανόνες επιστοποίησης και για να μπορέσουμε να είμαστε αυτόνομοι. Είχε λόγο ε, η ανάπτυξη του προγράμματος Γαλιλαίος. Θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο και σε ό,τι αφορά την άμυνα και πραγματικά χαιρετίζω τη δράση του Προέδρου Νταζάν ε, σχετικά με τα όσα έκανε στον τομέα της έρευνας. Πραγματικά αναρωτιέμαι αν θα πρέπει να υπάρχει μια ε, καλύτερη ε, συμφωνία και συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλίων αλλά και αν θα πρέπει να έχει αυξημένο ρόλο η Ευρωπαϊκή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας. Άκουσα την πρόταση για τον κοινωνικό σκέλος. Πραγματικά πώς μπορέσαμε, πώς δεν, πώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο για να υπάρξει η σύγκληση μεγαλύτερη. Η πολιτική συμφωνία στη Γερμανία είναι ένα πολύ καλό νέο. Θα πρέπει να υπάρχει αυτό το βαθμολόγιο έτσι ώστε η, ε, να υπάρξει η πολιτική βούληση να τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά. Ευχαριστούμε Ζαμπιέρ. Για δύο λεπτά τώρα το λόγο έχει η συνάδελφος Φερέιρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου πρέπει να ολοκληρώσει μερικά πράγματα. Πρέπει να κάνει αποφασιστικά βήματα. Η ενιαία εποπτεία των χωρών που συμμετέχουν είναι κάτι θεμελιώδες. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο ενιαίο Ταμείο Εξυγένσης με ενιαίους κανόνες για να μην χάνουν χρήματα οι αποταμιευτές και να χρηματοδοτούν οι τράπεζες στο ταμείο αυτό ανάλογα με το βαθμό κινδύνου που ελοχεύει στην κατάστασή τους. Πρέπει να σεβαστούμε την αρχή της αναλογικότητας. Η περίοδος είναι βέβαια δύσκολη για να ζητήσουμε από τους πολίτες να κάνουν περισσότερα, να δείξουν περισσότερη εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Η διακυβερνητική μέθοδος δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργήσε για να επιληθεί το θέμα του δημοσίου χρέους. Δεν λειτουργήσε με τις συμβατικές ρυθμίσεις του Συμβουλίου. Και έτσι, σε τέτοιους καιρούς δεν μπορούμε να δεχτούμε οι χώρες μέλη να αποφασίζουν για το μέλλον ε, των τραπεζών. Θα υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων, είναι προφανές. Το δεύτερο μάθημα που πρέπει να πάρουμε είναι ότι είναι οι τράπεζες οι οποίες πρέπει να πληρώσουν για την εξυγίανσή τους. Με ένα ισχυρό ταμείο λοιπόν, με συγκεκριμένες πιστοτικές γραμμές για να μπορέσει το ταμείο αυτό να λειτουργήσει με το που θα τεθεί σε ισχύ. Έπειτα λείπει ο τρίτος πυλώνας οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση με ενιαία εποπτεία, με ενιαίο ταμείο εξυγένσης, αλλά χωρίς ενιαίες εγγυήσεις όσον αφορά τις καταθέσεις. Αυτό είναι που λείπει, η εγγύηση καταθέσεων. Οι Ηνωμένε Πολιτείες το επέλεξαν για να οργανώσουν ε, την κατάσταση εκεί και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και δημιούργησαν μια ομοσπονδιακή υπηρεσία καταθέσεων. Οι αρμοδιότητες, οι αρμοδιότητες του οργάνου αυτού επίσης ενισχύθηκαν για να ανταποκριθούν στην κρίση του 2008. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο. Είναι σημαντικό το Συμβούλιο να διασφαλίσει την τραπεζική αυτή ένωση έτσι ώστε να μην επιδεινωθούν οι οικονομικές ανισορροπίες ή οι πολιτικές ανισορροπίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην ενισχύσουν Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπρόντς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η Επιτροπή θέλει περισσότερο ανταγωνισμό ενίας αγοράς για τους εξοπλισμούς, για τις αγορές εξοπλισμών, γιατί ε, οι κατακαιρματισμένες αγορές δημιουργούν προς τώρα γραφειοκρατία και κόστος. Όχι, δεν είναι το κατακαιρματισμένο των αγορών, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση που προξενεί περισσότερη γραφειοκρατία και κόστο. Βεβαίω, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι η τραγική ηρωνία, θα μπορούσε να αξιοποιήσει ε, όπως έχει κάνει άλλωστε και η Πολωνία και μπράβο της, ε, το σύστημα των πληστηριασμών όπως το προβλέπει η συνθήκη της Ευρωπαϊκής, για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε καθήκον να υπερασπιζόμαστε το εθνικό συμφέρον και η άμυνα έχει ζωτική σημασία για τα εθνικά συμφέροντα. Δεν μπορεί να αφαιθεί λοιπόν στο ελεύθερο ανταγωνισμό. Βεβαίως μπορεί να φαίνεται αδιανόητος ένας άλλος ευρωπαϊκός, ενδοευρωπαϊκός πόλεμος, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ε, προστασία μας, την ασφαλειά μας, την άμυνά Μην ξεχνάμε ότι η Βρετανία χρειάστηκε να πολεμήσει κατά τη επιθετική στάση και δράση των Αργεντινών. Ευχαριστούμε για δύο λεπτά ο Αντιπρόεδρος Προτασιέβιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει σημαντικά θέματα να συζητήσει συμπεριλαμβανομένης ε, και της βελτίωσης λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, αλλά και θεμάτων της πολιτικής άμυνας και ασφαλείας. Υπό το φως όμως των ε, εξελίξεων στο Κίεβο τις τελευταίες εβδομάδες και ιδιαίτερα τη τελευταία νύχτα, πιστεύω ότι πρέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της Ουκρανίας και των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτήν η απόφαση να μην υπογράψει συμφωνία σύνδεσης, απόφαση που ελήφθη την παραμονή της, της ε, της Συνόδου Κορυφής του Βίλνιους, είναι, ήταν πάρα πολύ δυσάρεστη. Αυτό όμως που συνέβησαν αυτή τη νύχτα με τις επεμβάσεις ε, της βίαιης καταστολής από τις αστυνομικέ δυνάμεις ειρηνικών διαδηλωτών και μάλιστα κατά τη στιγμή όπου είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική βρίσκεται στο Κίεβο ε, είναι αδύνατον να δικαιολογηθεί. Είναι ακατανόητη, δεν μπορώ να τη συγχωρήσω. Σήμερα, εδώ στο Στρασβούργο, την προσεχή εβδομάδα στις Βρυξέλλες, οφείλουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς τους χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που βρίσκονται στο Μαϊντάν, την ε, ε, πλατεία ανεξαρτησίας του Κιέβου, για να τους πούμε ότι είμαστε στο πλευρό τους, ότι τους στηρίζουμε, ότι δεν θα δεχθούμε ποτέ την άσκηση βίας σε μια χώρα η οποία επιδιώκει συμφωνία σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η βία δεν είναι ποτέ λύση. Και ως εκ τούτου προτείνουμε μια προφορική τροπολογία ε, για το ψήφισμα ε, το σχετικό με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Συνοδοκορυφή, ώστε να ασχοληθεί ιδιαίτερα με την Ουκρανία. Ευχαριστούμε. Για 1,5 λεπτό έχει τώρα το λόγο η κυρία Κλέβα Κέκους. Ευχαριστώ. Το προηγούμενο Μάιο συζητήσαμε για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και μιλήσαμε και για τα 30 συγκεκριμένα μέτρα που πρότεινε το Κοινοβούλιο. Μετά από μερικές ε, μέρες το Συμβούλιο κατέληξε σε ορισμένες αποφάσεις που αφορούσαν μία οπή χιλίων δισεκατομμυρίων. Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει αυτή την οδηγία μέχρι το τέλος του χρόνου και με αυτόν τον τρόπο να αρθεί το τραπεζικό απόρριτο. Σήμερα διαπιστώνω ότι στην ημερησία διάταξη της συνάντησης επόμενης εβδομάδας δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Φαίνεται ότι οι εκπρόσωποι των χωρών μελών είναι διατεθειμένοι να δώσουν πάρα πολλές υποσχέσεις και σε ό,τι αφορά τους G20. Όταν όμως τίθεται το θέμα των νομοθετημάτων δεν γίνεται απολύτως τίποτα δημοσιονομική οπή που υπάρχει υπονομεύει την εμπιστοσύνη στα οικονομικά συστήματα και μας στερεί πόρους για δημόσιες επενδύσεις. Η προβληματική της φοροδιαφυγής και φορολογικής απάτης θα πρέπει να είναι βασικό θέμα του Ευρωπαϊκού Εξάμεινου. Θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένοι στόχοι έτσι ώστε οι χώρες μέλη να συμπεριλάβουν στην ημερησία διάταξη το θέμα αυτό και να εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό τώρα. Έχει το λόγο η κυρία Μαρίν Λεπέν. Ευχαριστώ. Η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων αποδεικνύει τον κινησμό και την τρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αντιμετωπίζουμε κοινωνικό ντάμπινγκ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα αυτός ήταν και ο διπλός σας στόχος. Και να πέσουν οι μισθοί και να καταρρεύσει το σύστημα κοινωνικής προστασίας ε, στις πιο πρεγμένες χώρες. Κοινωνικά λοιπόν ε, γίνεται μια ευθυγράμμιση αλλά προς τα κάτω. Και εκλογικοί λόγοι ήταν να λένε όλοι «Α, κερδίσαμε, μπράβο, πολύ ωραία, συμφώνησαν» να αγωνιστούν, αλλά γιατί νομίζετε ότι όλα αυτά είναι κάτι καινούριο. Η ουσία της οδηγίας όμως που είναι καταστροφική και η οποία οδηγεί σε περισσότερη ενέργεια, σε περισσότερο ανταγωνισμό μέσα στον ίδιο χώρο ανάμεσα στις επιχειρήσεις, η επιθετική πολιτική μερικών χωρών που αποφελούνται από το σύστημα για να επιτεθούν στους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους. Πιστεύετε ότι οι εκλογείς θα δεχτούν να υπάρχει προτίμηση ε, προς τους ξένους αντί προς τους Γάλλους στη χώρα μου για παράδειγμα. Είναι δυνατόν. Τέλος, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η Ευρώπη σας είναι ο πόλεμος, ο οικονομικός πόλεμος και ο κοινωνικός πόλεμος. Ευχαριστούμε κυρία Λεπέν. Κυρία Γιακονσάλη. Θέλει να ρωτήσει κάτι κυρία Λεπέν. Κυρία Λεπέν δέχεστε για 30 δευτερόλεπτα. Ε? Ναι, σας ε, ευχαριστώ. Κύριε Λεπέν. Κύριε Λεπέν, δεν έχετε καταλάβει την ουσία της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων. Η ιδέα είναι ακριβώς να πληρώνονται τα ίδια χρήματα, οι ίδιες αποδοχές τους εργαζόμενους όπου και αν είναι αυτοί. Οπότε πώς είναι να τραβελώνετε έτσι το νόημα της οδηγίας αυτής. Ναι, κύριε Λεπέν, μα οι γαλλικές επιχειρήσεις νομίζετε ότι είναι ανόητες και οι ευρωπαίοι εκλογές είναι ηλίθιοι. Μα είδαν ποιες είναι οι συνέπειες της οδηγίας αυτής. Ναι, οι ίδιοι μισθοί βεβαίως, αλλά κοινωνικά βάρη που έχουν να κάνουν με τη χώρα προέλευσης. Οπότε η συνέπεια της απόφασης αυτής είναι 40.000 θέσεις απασχόλησης που χάθηκαν. Χάθηκαν στον οικοδομικό τομέα. Αν έχετε κάτι να πείτε, να σηκώσετε κι εσεί ε, την μπλε σα κάρτα, έτσι. Λοιπόν, έλεγα, 40.000 θέσει απασχόληση χάθηκαν στον οικονομικό τομέα. Και βέβαια και υπάρχει προτίμηση για του ξένου, γιατί σήμερα είναι υποχρεωμένε επιχειρήσει για να είναι ανταγωνιστικέ να ζητάνε απασχολούμενους από άλλε χώρε, εκεί όπου υπάρχουν ε, βάρη πολύ λιγότερα από εκείνα που υπάρχουν στι χώρε που εφαρμόζεται μια πραγματική κοινωνική προστασία, όπω για παράδειγμα η Γαλλία. Πρόεδρο, 30 δευτερόλεπτα έτσι κι αλλιώ είχατε στη διάθεσή σα. Υπενθυμίζω στου συναδέρφου μία μπλε κάρτα αναπαράμβαση επιτρέπεται. Για δύο λεπτά τώρα το λόγο έχει ο κύριος Δεγράντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι μεγάλες προσπάθειες και οι θυσίες που γίνονται για να διατηρηθούν σε γη κατάσταση τα δημοσιονομικά μας τα δύο τελευταία χρόνια αποφέρουν καρπούς. Όμως η ανάκαμψη ακόμα είναι εύθραυστη. Εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες. Κατά τη γνώμη μας, για να βγούμε από την κρίση, πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και να δούμε δύο πράγματα. Διαφοροποιημένη φορολογική πολιτική που να ενισχύει την ανάπτυξη. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που να οδηγήσουν στο να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί και να δημιουργήσουν νέε θέσει απασχόλησης. Μεταρρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα και στην Τραπεζική Ένωση στην εσωτερική αγορά. Επ' αυτού θέλω να πω, παρά τα όσα άκουσα, ότι οι συμφωνίες στις οποίες έχουμε οδηγηθεί μας δημιουργούν ελπίδα. Πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους και το Ταμείο για την Απασχόληση των Νέων ήδη φέρνει κάποια αποτελέσματα για την ισχύ των μικρομεσαίε επιχειρήσει. Το Ευρωπαϊκό αυτό Συμβούλιο πρέπει να οδηγηθεί σε μία απόφαση για την ανάκαμψη. Τραπεζική Ένωση. Επίγει, κυρίε και κύριοι, ενίο ταμείο εξυγίανση. Ενία αρχή δηλαδή. Επίση, που να το επιβλέπει η Επιτροπή το Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίση θα μπει σε βάθο όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Δεν μπορούμε να έχουμε καλή εξωτερική πολιτική αν δεν έχουμε αναπτύξει και κάποιες ικανότητες στον τομέα αυτό. Χρειάζεται ε, ισχυρή ηγεσία έτσι ώστε να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας και στη συνέχεια να κατανείμουμε τις αρμοδιότητες. Να μην υπάρχουν επικαλύψεις, να μην υπάρχουν αδυναμίες και να συμπληρωματικότητα των δράσεων αυτών, των στρατιωτικών και των μη στρατιωτικών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορούμε να αντιδρούμε καλύτερα, πιο αποτελεσματικά, πιο αποδοτικά, με περισσότερη ορατότητα. Και έτσι ενισχύεται και η εξοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που προσφέρει ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Λουί. Τώρα το λόγο έχει για δύο λεπτά η κυρία Περβάνς Μπέρες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε την Πρόεδρε τη Επιτροπής, ακούσατε ότι το Κοινοβούλιο δεν θέλει αυτές τις συμβάσεις. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι συμβάσεις είναι ένα είδος soft τρόικα που θα επιβάλλουν μεταρρυθμίσεις που θα πλήξουν πολλές χώρες μέλη. Από την άλλη το Συμβούλιο μας λέει ότι ενδεχομένως κάποια μέρα θα υπάρξουν κίνητρα. Εμείς δεν το πιστεύουμε. Θέλουμε να γίνουν και τα δύο παράλληλα. Σε ό,τι αφορά το ψήφισμα για τις τράπεζες, θα ήθελα να πω ότι το Κοινοβούλιο αυτό τη γνωρίζει ότι σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική αλληλεγγύη χρειαζόμαστε την κοινωτική μέθοδο. Με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας θελήσατε μια διακυβερνητική λύση. Αυτό δεν είναι ο δρόμος που θέλουμε. Δεν είναι η οδό που θα επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να κάνει κάτι με το σημειαίο σύστημα εποπτείας. Κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου, ακούστε με. Σε ό,τι αφορά την κοινωνική διάσταση, μήπως μπορείτε να με ακούσετε. Μήπως μπορείτε να με ακούσετε παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά την κοινωνική διάσταση, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει η εντολή του προκατόχου σας έτσι ώστε το θέμα της κοινωνικής διάστασης να συμπεριληφθεί. Ζητήσατε από την Επιτροπή να υποβάλει ένα ανακοινοθέν. Το ανακοινοθέν υπάρχει. Ε, λέτε ότι θα πρέπει να υπάρξουν δείκτες. Εμείς Λέμε ότι θα πρέπει να ενταχθούν στη διαδικασία, αλλά θα πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε γιατί εσείς λέτε αυτό που λέει η Eurostat. 125 εκατομμύρια άτομα απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια. Το 1 τέταρτο του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τη μοσονομική διάσταση, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τη συνάδελφο Κλεβάκεβου σε αυτό το τομέα να μένουμε αποτελέσματα. Και ελπίζω ότι οι εξελίξεις στο Λουξεμβούργο θα μας επιτρέψουν σοβαρά να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αναθεώρηση τη οδηγία για την αποταμίευση. Διαφορετικά θα διαπιστώσουμε ότι λείπουν χίλια δισεκατομμύρια ευρώ από τον προπολογισμό μα. Ευχαριστούμε Περβάν. για δύο λεπτά τώρα. Έχει το λόγο η κυρία Παλπέλτ. Κύριε Πρόεδρε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την οικονομία διαπιστώνουμε ήδη θετικά μηνύματα. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μπει στο σωστό δρόμο. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει, κύριε Επίτροπε, ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαναπάβεται και να θεωρεί ότι είναι ικανοποιημένη. Είχε έρθει η ώρα τώρα να αξιολογήσουν βεβαίω τα επιτεύγματα, αλλά και να δούμε εάν προκύπτουν ω αποτέλεσμα της διαχείρισης της κρίσης από πλευρά σας ή ε, εάν ε, είναι η ανεξάρτητη δράση και οι επιλογές των κυβερνήσεων των κρατών μελών εξίσου σημαντικές και αν θα πρέπει να τα κρίνουμε όλα στο πλαίσιο της ε, επικουρικότητας. Είναι σημαντικά λοιπόν ε, τα θέματα του Συμβουλίου. Σε ένα πράγμα όμως θέλω να υπογραμμίσω ότι πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται η, Ουκραίν, η Ουκρανία και να επιδειχθεί αλληλεγγύη με τους διαδηλωτές που βρίσκονται στους δρόμους από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να υιοθετήσουν τις δικές μας αξίες και αρχές γι' αυτό αγωνίζονται. Η εντολή μας λοιπόν έχει να κάνει με τα όσα έχουμε προσδιορίσει στην έκθεση η, το κατακαιρματισμό δηλαδή της οικονομικής αγοράς και τις ε, διαφορές, τα χάσματα που θα πρέπει να καλυφθούν. Η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν πρέπει να την παραγνωρίσουμε, αλλά δεν μπορούμε και να λησμονούμε. Και σε αυτό θα ήθελα να επισύρω την προσοχή του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ε, πρέπει να με επαγγελθούμε λοιπόν ώστε να μην εισαχθεί περιττή και ε, βαριά γραφειοκρατία. Επίσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις ε, προσπάθειες μέχρι τώρα των κρατών και οι ε, αξιολογήσεις, οι δικές αξιολογήσεις ανακράτος πρέπει να αναθεωρηθούν για να αξιολογηθεί και να ενισχυθεί ενδεχομένω συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Τα Εθνικά Κοινοβούλια επίση θα πρέπει να συμμετάσχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστούμε. Για 1,5 λεπτό τώρα, κύριο Σούντο Μπούλμαν. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, αν διαρωτηθούμε σήμερα ποια κατεύθυνση ακολουθεί ή μάλλον πια, ε, ποιο όργανο αυτό το οποίο παραεμποδίζει περισσότερο την οικονομική ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επάντηση είναι μία και σαφή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, Πρόκειται για το χώρο αυτόν ο οποίος δεν προσδιορίζει καμία σαφή πολιτική. Πρόκειται για το χώρο αυτόν ο οποίος δεν προσδιορίζει καμία ε, αλλαγή πορεία σε σχέση με τα λάθη που έχει ο ίδιος διαπράξει. Πρόκειται για το χώρο στον οποίο υποτίθεται ότι διαγράφεται πολιτική, μια ψεύδο πολιτική, χωρίς όμως να αναμβάνονται και οι πολιτικές ευθύνες για τα μέτρα τα οποία εισάγει. Είσαστε ε, εσείς που ζητάτε αυτή τη συμβασιακή συμβατική σχέση Προσπαθείτε δηλαδή πίσω από αυτή να, να Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας συντρέχει βέβαια σε αυτό, αλλά πρέπει να πείτε ποιος από ποιον, με ποιανού τα χρήματα θα καλύπτει τις ανάγκες σε κινήτρα οικονομικά, ποιος θα γράφει τα προγράμματα και πού, πού θα κρύβεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος αυτών των προγραμμάτων. Αυτό προσπαθείτε δηλαδή να δημιουργήσετε οδηγεί και αποκλειστικά οδηγεί στην ε, ε, οργάνωση μια νέα, μιας νέας πολιτικής τρόικας μιας αποτυχημένης πολιτικής δηλαδή την οποία προσπαθείτε να διευρύνετε χωρίς να ε, καταλάβετε τίποτα από την ανισόρροπη τελείως ακραία λιμπεραλιστική, ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική της Τρόικας. Είναι σαν να νομίζετε ότι εσείς κρατάτε την παγκέτα και διευθύνετε ενώ παίζει τη μουσική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο χορεύει στον ρυθμό της πολιτικής που θέλετε να υπαγορέψετε. Όχι, δεν δουλεύει αυτό. Το Κοινοβούλιο θέλει άλλη πολιτική. Ευχαριστούμε, κυρία Άρντε έχει μια ερώτηση. Δέχεστε. Παρακαλώ, Ρεβέκα Χάρμ. Για 30 δευτερόλεπτα όμως, έτσι. Ευχαριστώ και εγώ συμφωνώ με, την, ε, με τις επικρίσεις ε, που εξέφρασε ο κύριος Μπούλμαν, ο Σάρφος Μπούλμαν, 100% ε, ανακοίνωσε άλλωστε τις προθέσεις κυρία Μέρκελ πριν από μερικέ μέρε ένα επίσημο γεύμα. Ερωτώ λοιπόν ω κομμάτι του κυβερνητικού συνασπισμού οι σοσιαλιστέ συνάδελφοι του S5 τι σκοπεύουν να κάνουν σε σχέση με την Άγγελα Μέρκελ που τοποθετείται όπως τοποθετείται. Πολύ ευχαριστώ, λέει ο κύριο Πούλμαν. Θα απαντήσω στην ερώτηση της κυρία Χάρμ. Ρεβέκα. Γιατί νομίζετε ότι ξέρω τόσο καλά αυτά τα πράγματα, ακριβώς γιατί είχα την δυνατότητα να συζητήσω εντατικά το θέμα αυτό με την κυρία Μέρκελ. Εμείς πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό πρέπει να, η νέα όποια πολιτική πρέπει να υπαχθεί στον δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου. Το είπαμε και πριν από τις διαπραγματεύσεις και κατά τις διαπραγματεύσεις και μετά τις διαπραγματεύσεις για το συνασπισμό και πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει απαντήσεις γιατί δεν μας λέει ξεκάθαρα ε, το, τι μπορεί να γίνει μέσα στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια πολιτική μη δημοκρατική και στη διαδικασία αυτή θα αγωνιστούμε με όλους τους εμπλεκομένους για να οργανώσουμε το δημοκρατικό έλεγχο όπως πρέπει. Αυτή είναι η θέση μου, αυτή είναι η θέση της ομάδας του S5. Είναι η θέση εν γέννη των σοσιαλδημοκρατών. Και είναι γνωστό αυτό. Ευχαριστούμε εδώ. Για δύο λεπτά τώρα έχει το λόγο ο Πάολο Ραγγέλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι απαραίτητο η Ευρώπη να έχει της μια πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Αποτελεσματική. Πρέπει να έχει την, ε, την πολιτική αυτή λοιπόν στη διάθεσή τη. αλλά αυτό δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα βλέπουμε την κρίση στη Συρία, τη Λιβύη, τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη διχασμένα παρουσιάζουν διαφορετικέ το καθένα θέσει ενώπιον τη διεθνού κοινότητα. Πρέπει να ενισχυθεί λοιπόν αυτή η πολιτική για την Ευρώπη, διότι θα μα επιτρέψει να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία, να ενισχύσουμε αυτή τη διαδικασία της συνοχής σε συγκεκριμένους τομείς ότι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί δεν υπάρχει μια ισχυρή μονάδα πολιτικής προστασίας για την περίπτωση των φυσικών καταστροφών, ε, πυρκαγιές, ε, σεισμοί, καταποντισμοί, πλημμύρες, γιατί να μην υπάρχει μια τέτοια μονάδα πολιτικής προστασίας κοινή. Και γιατί στους τομείς αυτούς να μην υπάρχουν ήδη δυνατότητες για ανάπτυξη μιας έννοιας, μιας πρώτης έννοιας και ιδέας κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Αυτό βεβαίως θα πρέπει να τα προωθήσουμε ε, σε συνεργασία με τους Αμερικανούς εταίρους μας. Δεν είναι τυχαίο το ότι μας πιέζουν να επενδύσουμε περισσότερο στην άμυνα και την ασφάλεια, γιατί εκείνοι έχουν και άλλα μελήματα να, ε, που τους απασχολούν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να επενδύσουμε και εμείς από πλευρά μας και να δημιουργήσουμε μια πραγματική πολιτική της άμυνας. Και επίσης πρέπει να ωφεληθούμε από τις φυστάμενες υποδομές, ε, αγγλικό και γαλλικό πάνω απ' όλα δυναμικό που υπάρχει αξιοποιείται και μάλιστα θα αναφερθώ στην παρέμβαση στο Μάλι, στην επέμβαση στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, τις δυνατότητες για χρηματοδότηση αυτών των ε, προσπαθειών. Αυτά τα μικρά δηλαδή βήματα, τα οποία θα μας επιτρέψουν πιστεύω να δημιουργήσουμε μια πραγματική πολιτική της άμυνας. Ευχαριστώ Παόλο. Ένα μισή λεπτό, κυρία Βίλματ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Με χαρά βλέπω ότι η οικονομική και η κοινωνική πολιτική συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου. Ελπίζω πλέον να κάτσουν να συζητήσουν οι αρχικοί και κυβερνήσεων τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για να βελτιωθούν και να ενισχυθούν τα κοινωνικά και ε, οικονομικά δικαιώματα των πολιτών μας. Αλλά τι θα κάνουμε σε σχέση με την οδηγία για την απόσπαση. Είναι όλο και μεγαλύτερα τα παραθυράκια που ανοίγουν στην οδηγία αυτή, κυρίως και λόγω των ε, δυστυχώς ε, μη χρήσιμων, μη ωφέλιμων αποφάσεων του δικαστηρίου. Επιδεινώνεται λοιπόν το επίπεδο των προδιαγραφών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας. Πρέπει επιτέλους να δείξουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να καταδικάσουμε και να απαγορεύσουμε το κοινωνικό ε, dumping σε ένα σύστημα εργασίας ισότιμο και δίκαιο για όλους. Δυστυχώ, όμως τα άρθρα 9 και 12 των προτάσεων του Συμβουλίου επιδεινώνουν την κατάσταση την ασφάλεια δικαίου και ε, δεν επιτρέπουν διαφάνεια στην αλυσίδα της υπεργολαβίας. Είναι δυσάρεστες, δυσανάλογες και αναποτελεσματικές. Γι' αυτό επιτρέψτε μου με τον κινησμό που μπορώ ενδεχομένω να εκφράσω να πω ότι δεν περιμένω πολλά από το προσεχές συμβούλιο προτάσεις για τις ε, θέσεις εργασίας, για την φορολογία, για την ανάπτυξη μπορεί να φαίνονται εθελκτικές, αλλά το Συμβούλιο ακόμα δεν έχει πάρει θεραλές αποφάσεις. Μας, μας χρειάζονται λοιπόν πράξεις και όχι ρητορικέ. Η φίλη δύο, δύο λεπτά. Είναι γεγονός ότι η ατζέντα αυτού του Συμβουλίου έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πέρα από την Οικονομική και Νομισματική Ένωση την οικονομική και κοινωνική πολιτική αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το ζήτημα της άμυνας και ασφάλειας. δέκα χρόνια μετά τις πρώτες κινήσεις σήμερα η ατζέντα περιλαμβάνει πρώτον το στοιχείο της αξιολόγησης για το ποια είναι πραγματικά η επιτυχία και η απήχηση της μέχρι σήμερα κοινή και ε, ε, αμυντικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας δεύτερον πώς αναπτύσσονται οι αμυντικές ικανότητες και τρίτον τι γίνεται με τις αμυντικές βιομηχανίες. Όσο αφορά στην αξιολόγηση υπάρχει ήδη ένα κείμενο της ε, υπάτης εκπροσώπου το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον αλλά και μια σειρά εκθέσεων του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου τα οποία το συμβούλιο οφείλει να χρησιμοποιήσει τα κείμενα αυτά τα οποία δείχνουν την κατεύθυνση. ακόμα και αν βρισκόμαστε σε εποχή δημοσιονομικής κρίσης μπορούμε κάλλιστα με λιγότερα χρήματα να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα αν συνεργαστούμε όπως πρέπει αν λειτουργήσουν σωστά τα eu battle groups αν λειτουργήσει σωστά το πρόγραμμα ατένα αν πραγματικά στην αμυντική βιομηχανία ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία και όχι μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και τις μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διάφορες χώρες και μπορούν να συμβάλλουν στην παραγωγή οπλικών συστημάτων στην ερώτηση αν σε μια εποχή κρίσης με τόση ανεργία εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με την αμυντική πολιτική ναι γιατί αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε στην καρδιά της ύπαρξης μιας πιο ενιαίας ευρώπης είναι μείζον πολιτικό θέμα και από την άλλη πλευρά μπορούμε κάλλιστα μέσα από τα δημοσιονομικά μέτρα να ικανοποιήσουμε τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις να δώσουμε περισσότερη ασφάλεια στον ευρωπαίο πολίτη και περισσότερη αυτοπεποίθηση κύριε πρόεδρε σε σχέση με το τι είναι και τι αισθάνεται πως είναι η ευρώπη. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γεννάκου. Ένα μισή λεπτό. Ο κύριος Λόμπεθ Αγγελά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελεί πάντοτε πολιτική συνάντηση ύψης του επίπεδο. Εδώ μιλήσαμε για τις σκέψεις μας που θα επικεντρωθούν στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα, την αδότα άμυνας και τον τομέα βιομηχανίας, τον αμυντικό της Ευρώπης. Ο κύριος λόγος όμως και η κύρια ανησυχία είναι οικονομική. Οι περικοπές που μας ε, επιβάλλουν να βελτιστοποιήσουμε τις πολιτικές αυτές τις χώρες μέλη μας οδηγούν να πούμε ότι περιμένουμε ότι έχουμε προσδοκίες αντίστοιχες με αυτές που έχουμε την Τραπεζική Ένωση. Δεν φτάνει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό εποπτείας και εγγύηση των καταθέσεων. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις αρμοδιότητες της Κομισιόν στη διαχείριση αυτού των νέων συστημάτων Τραπεζικής Ένωσης, αλλά και αυτού του ελέγχου που θα πρέπει να ασκεί το, κοινο, το Κοινοβούλιο. Και όλο αυτό γιατί πλησιάζουν οι ευρωεκλογέ και είναι εύκολο να αφαιρεθούμε. Το 2014 λοιπόν θα δούμε ότι θα έχουμε από τη μια μεριά τους ευρωπαϊστές και την ανάπτυξη που δείχνουν πολλές έρευνε και την αύξηση ευρωφοβικών και αντιευρωπαϊκών στάσεων. Οι ευρωεκλογέ λοιπόν θα αποτελέσουν μια τελευταία ευκαιρία για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε την οικονομική πολιτική που επέβαλε αυτέ τι περικοπέ, που οδήγησε την αμυντική μηχανία τη Ευρώπη στη χειρότερη στιγμή τη ιστορία τη. Και θα πρέπει βεβαίω να προωθήσουμε την κοινωνική ατζέντα και την δημιουργία απασχόληση. Ευχαριστώ, Φερνάντο, Πρόεδρο. Ε, Υπάρχει μια συνάδελφος η Κακαβάχη η οποία θέλει να κάνει μια ερώτηση. Φερνάντο, την αποδέχεσαι? Ναι ή όχι Φερνάντο, πες μου. Ναι, καλά. Κάριν, 30 δευτερόλεπτα. Στα πλαίσια του πακέτου για τις κοινωνικές επενδύσεις η Κομισιόν παρουσιάστηκε ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αυτά τα θέματα. Ε, δεν πιστεύεις ότι στα πλαίσια του εξοπλισμού και της άμυνας θα είχε νόημα η... να εξοπλιστούν οι Ευρωπαίοι κατά των ασθενειών. Ε, αυτό μπορεί να γίνει όμως μόνο με ένα στιβαρό σύστημα υγείας. Δεν πιστεύεις ότι με αυτή την επένδυση συμβάλλουμε στην ανάκαμψη εκτός από την υγεία των Ευρωπαίων και της οικονομίας μας. Ευχαριστώ Καρίν Φερνάντο. Θέλεις να απαντήσεις 30 δευτερόλεπτα κι εσύ. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση όμως απαιτεί να πούμε με σαφήνεια ότι δεν γίνεται να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια ότι κάνοντας περικοπές και υποχρεώντα τι χώρε μέλη να περικόψουν το κράτο πρόνοια, μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα την ευημερία και τα κοινωνικά δικαιώματα μαζί με το δικαίωμα για την υγεία και την πρόσβαση στη δημόσια υγεία την ποιοτική στι χώρε μέλη. Βεβαίω αυτό αφορά και την προσπάθεια προσέγγιση που κάνει η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλεια και Αμυνα, γιατί ακολουθεί δυστυχώ οικονομιστική προσέγγιση. Μα υποχρεώνουν οι περικοπέ να μειώσουμε την δυνατότητα άμυνα. Αλλά αυτό που θα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι το ευρωπαϊκό εγχείρημα το οποίο θα είναι κοινό και αποδεκτό από όλου. Ευχαριστώ. Ο κύριο δύο λεπτά. Καταρχήν για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι τα κράτη-μέλη που εφήρμοσαν πολιτική δαπανών ε, αντιμετώπισαν κρίση σε σχέση με αυτούς που επέλεξαν τις μεταρρυθμίσεις. Ε, είτε είναι έξω από την κρίση είτε σταδιακά ανακάμπτουν. Αυτό είναι σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όταν συζητάμε για το άνοιγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ελευθερία εγκατάστασης και απασχόλησης, αυτό δεν είναι απειλή. Αυτό είναι η ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολιτική ισχύ, αλλά και κάποιες θεμελιώδεις αξίες που πρέπει να διαφυλάξουμε. Τρίτον, η συζήτηση για τις πιο θεμελιώδεις και σημαντικές αξίες της δημοκρατίας, της σταθερότητας και της ειρήνης στην Ευρώπη ε, πρέπει να αναδείξει το γεγονός ότι τώρα σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε και να το σεβόμαστε γιατί ε, εκείνοι ζητούν την ελευθερία, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, διαφανείς κοινωνίες, διαδηλώνουν για όλα αυτά. Είναι λοιπόν μια εποχή μετασχηματισμού και πρέπει να ανταποκριθούμε. Δεν διαδηλώνουν παρά μόνο γι' αυτό, ενώ υπάρχουν άλλοι που εν θέλουν να κατησχίσουν άλλες δυνάμεις η Ουκρανία θα πρέπει να ε, συνάψει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ασκήθηκαν άλλες δυνάμεις σκοτεινές. Εμείς πρέπει να υποστηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι θα διαφυλάξουμε και την ευρωπαϊκή ειρήνη και τη σταθερότητα. Αν δεν ανταποκριθούμε σε αυτό πρέπει να συζητήσουμε για το πώς θα ε, διαμορφώσουμε καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Χέρτσο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εγχείρημα ειρηνευτικό και έτσι πρέπει να παραμείνει. Ε, οι ειρηνικές λύσεις είναι σημαντικές και η αλληλεγγύη προς τον Ουκρανικό λαό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δημοκρατικό έλλειμμα υπάρχει και στις δυτικές κοινωνίες και οικονομικό έλλειμμα σε πολλές από αυτές. Εκεί πρέπει να επιτελέσουμε πρόοδο. Σε ό,τι αφορά την αγορά στον τομέα της άμυνας, την Τραπεζική Ένωση, την οικονομική κοινή διακυβέρνηση, ε, όλα αυτά σημαίνουν ότι πρέπει να προσφέρουμε περισσότερη Ευρώπη. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στις Βρυξέλλες μιλούν για περισσότερη Ευρώπη, αλλά στις πατρίδες τους ασκείται περισσότερη κυρίαρχη εθνική πολιτική οι αρχηγοί των κυβερνήσεων θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση, να δεχτούμε ε, νέους ανθρώπους. Ε, αλλιώς ε, θα προχωρήσουμε σε αποκλεισμό αλλά και κατάρρευση. Ζητώ να είναι συνεπείς οι αρχηγοί των κυβερνήσεων και να εξηγήσουν αυτό που συμφωνήσαμε στις Βρυξέλλες, που συμφωνήθηκε στις Βρυξέλλες, να το εξηγήσουν στους λαούς τους. Ευχαριστώ, Δύο τώρα για τον κύριο Μίτσελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μερικές από τις σκέψεις μου για την ανάκαμψη και την ε, ανάπτυξη έχουν ήδη λεχθεί, αλλά θα ήθελα να μιλήσω ε, για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Έρχομαι από μια χώρα ουδέτερη από στρατιωτικής απόψεως ε, δεν ε, βεβαίως να παίρνουμε μαθήματα από το Sinn Féin ε, για τους πόρους γιατί χρυσάστηκε να, στην Ιρλανδία να πληρώσουμε πάρα πολλά για τις στρατιωτικούς πόρους από τα χρήματα των φορολογουμένων. Αλλά βεβαίως δεν αφαιρέθηκαν από το φορολογικό σύστημα και χρειάστηκε να τα χρησιμοποιήσουμε για στρατιωτικούς πόρους έχουμε την κληρονομιά αυτής της οργάνωσης και που θέλει τώρα να ξαναγράψει την ιστορία. Η Ιρλανδική οικονομία έχει παρόλο που έχει την, την, το Sinn Féin και τις καταστροφές του Sinn Féin έχει ανακάμψει και θα πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμής στην Ιρλανδική κυβέρνηση που έκανε το παν ε, για να μπορέσει να ανατάξει αυτή την οικονομία. Όσον αφορά την, πολιτική, την κοινή πολιτική ε, Άμυνα, μου φαίνεται ότι σε εποχές λιτότητας μια καλύτερος συντονισμός ανάμεσα στα 28 ε, κράτη-μέλη θα ήταν καλό αντί να έχουμε ξεχωριστούς προϋπολογισμούς αμυντικούς για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, να βοηθήσουμε τις πιο, τα πιο αδύναμα στρώματα του, της κοινωνίας, να υπάρξει αλληλεγγύη προς όλες τις κατευθύνσεις. Υπάρχουν βεβαίω τα θέματα κυριαρχίας που απασχολούν. Θα πρέπει να πούμε ότι για αυτούς που είναι ουδέτερες χώρες που δεν θέλουν κοινή πολιτική έχουμε βεβαίω ορισμένες δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ ε, και της Δυτικοευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είναι αυτόματες αυτές οι διατάξεις. Θα μπορούν οι χώρες να επιλέγουν και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε την ε, πρόπτικη να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την αλληλεγγύη στην κοινή άμυνα που είναι προς δύο κατευθύνσεις. Μερικές ουδέτερες χώρες ε, δεν έχουν φροντίσει για την άμυνα ε, της χώρας τους έχουν κοπεί οι δαπάνες. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις οικονομίες αυτές με τρόπο πιο αποτελεσματικό, να υπερασπιστούμε τις ανάγκες ε, των πολιτών μας και να έχουμε αυτή την συζήτηση με πολιτισμένο τρόπο. Ευχαριστώ Γκέι. Η κυρία Ναγκόμες για ένα λεπτό. Κοιτάξτε την Λαπεντούζα και κοιτάξτε την ανασφάλεια στη Λιβύη για να δούμε, σε, βρίσκεται σε βαθιά πολιτική κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορεί να συντονίσει, συντονίσει τις πράξεις και οι αντιζηλίες ανάμεσα στα κράτη-μέλη θέτουν την ασφάλεια σε κίνδυνο και ακόμα δημιουργούν μεγάλη ανθρωπιστική κρίση. Έχουμε θαλάσσιες απειλές, οργανωμένες τρομοκρατίες, εγκλήματα, που δεν καλύπτονται από το Συμβούλιο που παρά την ρητορική δεν ερευνά για τα θέματα βιομηχανίας και έρευνας για να έχουμε μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Στο αντίθετο, δείτε τη χώρα μου, την Πορτογαλία, ε, που ε, κλείνει τα ναυπηγεία. Δείτε ποια είναι η στρατηγική παραγωγή, ε, πώς έχουμε ε, την απειλή και δούμε, δείτε τι γίνεται από, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Θα δούμε ότι πώς περικόπτονται οι προϋπολογισμοί οι αμυντικοί. Έχουμε επίσης διάφορες δημόσιες συμβάσεις αμυντικές με διαφθορά και στρέφονται τα μέσα. Για δείτε το Μάλι, την ε, Κεντρική Αφρική, την ε, Γαλλία, μόνη της που δρά. Θέλετε περισσότερες αποδείξεις ότι το Συμβούλιο και η Κομισιόν αποτυγχάνουν στην πολιτική αυτή, αποτυγχάνουν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της Ευρώπης. Ευχαριστώ, Άννα. Δύο λεπτά. Ο κύριος Φρανκ Εγγέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι μόνο η ασφάλεια της Ευρώπης που απολύεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είμαι ακόμα και το δίκαιο που απειλείται ε, της Ευρώπης. Ας αρχίσω μιλώντας ε, για την Τραπεζική ε, Ένωση. Κανείς δεν πιστεύει στην Τραπεζική Ένωση. Αυτή η Τραπεζική Ένωση είναι εσωτερική ενδογενή στην κρίση και στην ανόητη πολιτική λιτότητα με την οποία μαστιγώνουμε τις χώρες μας. Ας τελειώσουμε, ας τελειώσουμε, αλλά ας ε, προβούμε ε, σε μια σχεδιασμό πολιτικών που να αξίζουν και που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Διότι εκεί, κύριε Πρόεδρε, διαπιστώνω ότι υπάρχουν εκτροπές από μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αρχίζω να θεωρώ ότι είναι προβληματικές και σαν σανδαλώδεις. Ο Πρωθυπουργό, ο Βρετανός, δημοσίευσε άρθρα για να νοθεύσει βία ε, το κράτος δικαίου το ευρωπαϊκό. Είναι ε, σαν να είχε ένα κράτος ανεξέλεγκτο χωρίς κοινωνική ασφάλεια ενώ τελικά πρόκειται μόνο για τη δυνατότητα για τους Ευρωπαίους να μπορούν να διασχίζουν ε, τα ευρωπαϊκά σύνορα για να μπορούν να εργαστούν και να υποφεληθούν από ορισμένε εγγύησει αλληλεγγύης. Ο Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι ο μόνος που έχει αυτή την αντίληψη, διότι υποτίθεται ότι έχει φίλους που θα ήθελαν μαζί του να περιορίσουν την ελευθερία ε, διακίνησης και κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι λυπηρό, λυπηρότατο και θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, που δεν είναι πιο, το πιο αποτελεσματικό και ευρωπαϊκό όργανο τουλάχιστον να είναι ικανό να ανακαλέσει στην τάξη τα μέλη που για λόγους λαϊκίστικους και ψηφοθυρικούς δεν διστάζουν ε, μπρος στην αμφισβήτηση των βασικών και κτημένων της, της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Ευχαριστώ Φρανκ. Δύο λεπτά. Ο κύριος ε, Κέλλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε μπορούμε να πούμε ότι η, μεγάλη, επόμενη μεγάλη κρίση στην Ευρώπη κατά πάσα πιθανότητα θα είναι κρίση ασφάλειας και άμυνας. Η γειτονιά μας έγινε πιο ασταθής και απρόβλεπτη προς όλες τις κατευθύνσεις ε, τρομοκρατικές απειλές, ε, κυβερνητικά εγκλήματα που εν μέρη ε, προωθούνται από κράτη ε, αυξάνονται. Όμως η μεγαλύτερη απειλή είναι η αδυναμία της Ένωσης να αντιδράσει σε όλα αυτά. Οι αμυντικοί προϋπολογισμοί ήταν τα πρώτα θύματα της λιτότητας. Ανησυχώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά δεν πόρεσε να αντιδράσει σε αυτό το δίλημα μεταξύ αυξημένων απειλών και μειωμένων αμυντικών δυνατοτήτων. Η συνένωση, ο επιμερισμός και η κοινή χρήση είναι ένα θέμα, αλλά μπορεί να δώσει απαντήσεις στη συνασφάλεια. Νομίζω ότι το πρώτο καθήκον του Συμβουλίου ε, είναι να σταματήσει τον εφησυχασμό και τη μειοπική προσέγγιση. Ο πρώτος στόχος μας είναι να ε, συγκεντρώσουμε την ε, στήριξη της κοινή γνώμης. Οι πολίτες εκτιμούν την ασφάλειά τους πάνω απ' όλα, αλλά δεν μπορεί αυτή να παρασχεθεί δωρεάν. Είναι μεγάλη η πρόκληση από άλλες χώρες που δαπανούν πάνω από 4% ε, για το σκοπό αυτό. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την Ρωσία έτσι η οποία ε, διεξάγει πολιτικό πόλεμο ενάντια στους γείτονες ε, που απείλησε την Γεωργία και που το στρατηγικό δόγμα της απειλεί τους γείτονες. Ε, πρέπει και εμείς να έχουμε αμυντική δυνατότητα. Αν η Ευρώπη δεν αναλάβει δράση, το Κρεμλίνο θα είναι ελεύθερο να προωθήσει τους στόχους του στην Ουκρανία, Μολδαβία και στις χώρες της Βαλτικής και στη Γεωργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Τούνε, τελευταία παρέμβαση σε αυτό το γύρο ο κύριος Κάρας, αντιπρόεδρος, για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχήν ε, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Πριν από ένα χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης. Αυτό κατέδειξε ότι το ειρηνευτικό εγχείρημα της Ευρώπης είναι επιτυχημένο. Έχουμε συνεργασία, ε, κατανόηση ε, ο ένας για τον άλλον. Μπορούμε μαζί να λύνουμε προβλήματα. Ε, απέναντι σε ποιον αμυνόμαστε. Απέναντι στον εαυτό μας. Τώρα οι αμυντικές προσπάθειες θα πρέπει να συνενωθούν ούτως ώστε να μπορούμε να επιλύουμε από κοινού προβλήματα εντός και εκτός της Ευρώπης. Η μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επ' αυτούς δείχνει ότι η συνένωση των δυνάμεων εδώ εξοικονομούν 130 δίσε το περισσότερο, 26 δίσε το λιγότερο και αυτό αυξάνει ταυτόχρονα και την αποτελεσματικότητά μας. Καλό τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να προχωρήσουν σε αύξηση της αποτελεσματικότητας με μείωση του κόστους. Δεύτερον, η Νομισματική Ένωση ε, προϋποθέτει οικονομική και κοινωνική ένωση, όχι με διμερείς συμφωνίες, αλλά με βάση το, το ενωσιακό δίκαιο, με δημοκρατική νομιμοποίηση και έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και η Τραπεζική Ένωση είναι η προϋπόθεση ώστε η τραπεζική εποπτεία να έχει επιτυχία θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση για την Τραπεζική Ένωση πριν από τις ευρωεκλογέ. Έτσι θα σηματοδοτήσουμε ότι είμαστε σοβαροί στην αντιμετώπιση της κρίσης. Ευχαριστώ, Τμάρ. Ολοκληρώσαμε τον γύρο ομιλητών που μίλησαν προσωπικά. Έχουμε κάποιους για το Catch και ξέρετε ότι στο λεπτό ακριβώς θα σας κόβω το λόγο. Θα μιλήσετε όμως όλοι Έστω και αν ήσασταν περισσότεροι από θα έπρεπε. Η κυρία Μαγκίνες καταρχάς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ το, την Κομισιόν και το Συμβούλιο για αυτή την συζήτηση. Επίτροπε, είπατε και ευχαριστώ που το αναγνωρίζετε ότι οι Ιρλανδοί ήταν επίμονοι και πολύ υπομονετικοί. Εμεί βγήκαμε από το πρόγραμμα Bailout, ήταν πολύ σκληρά αυτά τα τρία χρόνια. Θα ήθελα όμω να τονίσω ότι παρά κάποια σχόλια από συναδέλφου νωρίτερα, η Ιρλανδία παραμένει μια θετική είδηση. Να σας πω κάποιες από τις καλές ειδήσει. Έχουμε την επιστροφή της ανάπτυξης. Η οικονομία ξανακερδίζει ανταγωνιστικότητα. Οι εξαγωγές είναι στο μέγιστο ιστορικό και επέστρεψε η εμπιστοσύνη. Τα επιτόκια στα κρατικά ομόλογα έχουν πάει σε ανοιχτά επίπεδα. Αυτή η ανάκτηση για κάποιους οικονομική και η ανάκαμψη δεν είναι καλή γιατί προποθέτει μια πολιτική αποτυχία. Γι' αυτό είναι φοβερό να το πει κανεί εδώ στην Ολομέλεια. Ε, διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μαγκίνε. Ο κύριο Πάσκο έχει το λόγο. Νομίζω ότι πλησιάζει το Συμβούλιο για την Άμενα και δύο είναι οι λόγοι για του οποίου έχουμε υψηλέ προσδοκίε. Με την άμυνα δεν ασχοληθήκαμε από το 2008 και είναι η άμυνα ε, που ε, στην κρίση τώρα ε, έχει τις μεγαλύτερες περικοπές. Μπήκαμε σε μια εποχή όπου έχουμε φόβο να χάσουμε την, την ψήφο τη λαϊκή. Το θέμα ασφαλείας είναι σημαντικό. Έχουμε δυσκολίες αν έχουμε θελοντές. Η βιομηχανία χάνει εξειδικευμένο προσωπικό και τα όπλα μας είναι ξεπερασμένα. Η τεχνολογία έχει μειωθεί και ο αναδιόμενος κόσμος κόσμος βρίσκεται στο επίκεντρο του κόσμου. Για να μην περάσουμε το σημείο της μη επιστροφής δεν πρέπει να πάψουμε να περικόπτουμε τους προϋπολογισμούς και να αποδώσουμε σημασία στην άμυνα ε, στο επόμενο Συμβούλιο. Ευχαριστώ Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Χρυσόγελος, Νίκος. Για αυτά που αναφέρω μερικά παραδείγματα ε, για το ευρωπαϊκό εξάμεινο δεν μπορεί να βλέπουμε μόνο τους δείκτες μακροοικονομικούς αλλά πρέπει να συνδέουμε τους δείκτες αυτούς και με κοινωνικούς δείκτες. παράδειγμα η επίτευξη δημοσιονομικής εξυγίανσης δεν πρέπει να πλήττει την κοινωνική συνοχή. στην ελλάδα έχουμε πάνω από 28% ανεργία 60 64% ανεργία μεταξύ των νέων. ακόμα και αν πετυχαίναμε δημοσιονομική εξυγίανση θα ήταν σε βάρος της συνοχής κοινωνίας αλλά ούτε δημοσιονομική εξυγίανση πετυχαίνουμε η πολιτική λιτότητα είχε σαν αποτέλεσμα να καταστρέψει την παραγωγική βάση και την κοινωνική συνοχή αλλά δεν μείωσε το χρέο. η πρόσφατη έκθεση του οσα λέει ότι ό,τι πετύχαμε με το κούρεμα και με άλλα μέτρα για τη μείωση του χρέου, εξουδετερώθηκε από την αύξηση του ίδιου ποσοστού του χρέους δηλαδή μειώθηκε το χρέος 38,5% με το κούρεμα και λόγω τη ύφεση αυξήθηκε πάλι 38,5% δηλαδή δεν πετύχαμε τίποτα tiempo. Tiene la palabra el señor Murphy. Ευχαριστώ. Έχει το λόγο ο κύριος Ευχαριστώ. Ο Όρουελ το 1984 είπε ότι ε, λέμε σκόπιμα ε, ψεύδι και τα πιστεύουμε. Ε, δεν υπάρχει καλύτερος ε, ορισμός σχετικά με την ιστορία της Κομισιόν για την Ιρλανδική επιτυχία. Ε, επιστροφή κυριαρχίας. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά ε, στοιχεία τα οποία ε, ε, ε, περιορίζουν τον Ιρλανδικό λαό. Έχουμε και μετά το πρόγραμμα επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχουμε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, οι δέσμοι των δύο νομοθετημάτων, των έξι, περισσότερα συμφωνίες για τη λιτότητα. Έχουμε συνέχεια μια τρόικα σε όλη την Ευρώπη. Ε, η μάχη και ο αγώνας κατά του ιμπεριαλισμού θα μπορούσε και σήμερα να ισχύει. Όσο λιγότερα λέμε για την ορ... διακοπή. Τελειώσε ο χρόνος σας. Έχει το λόγο και ο Σικέρσκι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η κοινή πολιτική για την άμυνα και την ασφάλεια αποτελεί ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Απαιτεί να συνενέσουμε και να συμβάσουμε τα οικονομικά και τα πολιτικά συμφέροντα. Τα οικονομικά συμφέροντα εδώ είναι πολύ σημαντικά και τα εμπορικά συμφέροντα πολλές φορές ξεπερνούν και υπερβαίνουν τις αξίες μας. Η πλειοψηφία των ομιλητών αναφέρθηκε στην Ουκρανία. Όμως έχουμε κάποια αόριστη δήλωση και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάρα πολλές χώρες ε, τηρούν σιγή για αυτό το θέμα για να μην θίξουν τις σχέσεις με τη Ρωσία. Η κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας βασίζεται νομίζω σε κάποιες κοινές αξίες οι οποίες είναι βασικές για τη λειτουργία μας. Θα ήθελα να αφιστήσω λοιπόν την προσοχή σας στο γεγονό ότι η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ μεγάλη όταν έχουμε να κάνουμε με απειλή ανθρωπίνων ζώων. Ο κύριος Πίκουλα, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ο Μάνφρεντ Βέρνερ είπε ότι καμιά φορά τα πράγματα τα παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίζει τη δημοκρατία και εγώ προσωπικά θα ήθελα να υποστηρίξω τον τομέα της άμυνας της Ευρωπαϊκής. Η άμυνα νομίζω είναι απαραίτητη σήμερα και ε, παρουσιάζει και άλλες πτυχές, οικονομικές, κοινωνικές. Η σταθερότητα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό θα πρέπει μαζί από κοινού ως εταίροι να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε τις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κροατία συμμετέχει σε ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές ειρήνης και σήμερα βλέπουμε παγκοσμίω ότι είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε την άμυνα την ευρωπαϊκή. Γι' αυτό ακριβώ βλέπω θετικά το Συμβούλιο του Δεκέμβρη. Ευχαριστώ. Τελειώσατε το χρόνο σα, λέει ο Πρόεδρο. Έχει το λόγο τώρα ο φίλος Σον Κέλλη. Uh, Νομίζω ότι αυτό τη σύνοδο κορφής έχει μεγάλη σημασία στα 4,5 χρόνια που είμαι εδώ ο, ο καθηγητής Νότολ είπε ότι το ευρώ δεν κατέρευσε και δεν κατέρευσε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι το ευρώ είναι ασφαλές και έχουμε ανάκαμψη, επιστροφή στην ανάπτυξη και η χώρα μου θεωρείται ένα παράδειγμα επιτυχίας χάρη στην βοήθεια που λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλους. Αλλά θα πω ένα πράγμα το χρέος μας έχει ε, γίνει πάρα πολύ σημαντικό ε, που είναι κάτι το διπλό από ό,τι ε, προτείνεται στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας είχαν υποσχεθεί το 2012 ότι δεν θα έχουμε δεύτερο πρόγραμμα στήριξης, αλλά βλέπουμε ότι η Ιρλανδία είναι παράδειγμα επιτυχίας. Ευχαριστώ, Σον. Η κυρία Φλασικόβα Μπενόβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι από τα κυριότερα θέματα του Συμβουλίου Κορυφής θα είναι η οικονομική πολιτική. Είναι αναπόφευκτο να εμβαθύνουμε την νομισματική και οικονομική ένωση. Χρειαζόμαστε όμω την ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε περισσότερε θέσει εργασία, περισσότερη κοινωνική συνοχή. Η πιο μεγάλη προτεραιότητα είναι η υποστήριξη τη απασχόληση και η κοινωνική ευημερία. Ε, χρειαζόμαστε συστημικά μέτρα, φίλε και φίλοι, και όχι μόνο προσωρινά τα οποία μόνο οδηγούν σε αρνητικέ επιπτώσει στην απασχόληση. Ο κόσμο υποφέρει από την κρίση και υποφέρει εδώ και πολύ καιρό. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε και να ενισχύσουμε την χρηματοδότηση της οικονομίας. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις ε, επενδύσεις. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και θα πρέπει να αποτρέψουμε τις κοινωνικές ταραχές οι οποίες θα, προκαλέσουν, θα προκληθούν από τα μέτρα αυτά. Ευχαριστώ Μονίκα Λίγο Πρόεδρος. Ε, τέλειωσε ο χρόνος σου. Τελευταίος ομιλητής σε αυτό το γύρο, ο κ. Ρουσκέβικ. President, jeħtieġ li l istati membri jieħdu inizjattiva u b'sens ta' solidarjetà jagħtu sehemhom ε, σετικά με την αλληλεγγύη πρέπει να βρεθεί μια λύση για την μετανάστευση γύρω από την Μεσόγειο. Όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες απέναντι σε αυτή την πρόκληση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής να μπορέσει επίσης να προσπαθήσει να βρει ε, μηχανισμούς για το θέμα αυτό. Επίσης τα μέτρα ε, θα πρέπει να μετατραπούν σε συγκεκριμένες και αποτελεσματικές δράσεις. Η δυσανάλογη ευθύνη της Μάλτας μας δείχνει ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η πολιτική αυτή και το Δουβλίνο, η πολιτική του Δουβλίνου ε, για να υπάρξουν οι στόχοι της, του Στοκχόλμης, η ε, συνεργασία με χώρες μη μέλη για την μετανάστευση και το άσυλο είναι επίση σημαντικά. Ευχαριστώ Τζοζεφ. Ολοκληρώσαμε αυτό το γεμάτο γύρο ομιλητών. Μας μένουν τα σχόλια της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Καταρχάς, εξ ονομαστός του Συμβουλίου, θα δώσουμε τον λόγο, μάλλον θα μιλήσει, ο κύριος Σεύκοβης, ο Αντιπρόεδρο Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Uh, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τη συζήτηση. Θα προσπαθήσω σύντομα να αντιδράσω και να απαντήσω στα θέματα που έθεσαν ως επιτοπλίστων οι βουλευτές, ε, μηχανισμός, ε, ενιαίος μηχανισμός εξυγένσης Ουκρανία δημόσιες συμβάσεις. Ευχαριστώ για την ξεκάθαρη θέση σας για την Ουκρανία. Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι είμαστε στο πλευρό του Ουκρανικού λαού, στηρίζουμε το δικαίωμά τους να ακολουθήσουν το ευρωπαϊκό μονοπάτι και ευχαριστώ που καταδείξατε την αλληλεγγύη σας τόσο ξεκάθαρα. Συμφωνώ με τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων που ανέδειξαν το γεγονός ότι οι εικόνες από το Κίεβο, από την πλατεία μας θυμίζουν τη σημασία των ελευθεριών, των αξιών που έχουμε τόσο πολύ εγκολποθεί και τις θεωρούμε στην Ευρώπη δεδομένες. Ε, όπως ε, ε, είδαμε σήμερα το πρωί, όπως είπαμε σήμερα το πρωί, είναι πολύ σημαντικό να τις προασπίζουμε αυτές τις αξίες και ελευθερίες ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά αυτή είναι η συνεχιζόμενη μάχη ενάντια σε όλους αυτούς που θέλουν να περιορίσουν την ελευθερία διακίνησης, εργασίας, τα βασικά χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάνουν την Ένωσή μας τόσο μεγάλη. Οι ελευθερίες που ε, εκτιμούν τόσο οι πολίτες μας και είναι σαφές μας καθήκον να εργαστούμε εδώ όλοι μαζί και να δώσουμε μάχη για τις ελευθερίες αυτές και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για το θέμα της άμυνας θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμίσουμε σε κάποια αξιότιμα μέλη ότι η ΚΕΠΑ και η ανάπτυξή της έχει ήδη προβλεφθεί στη συνθήκη της Λισαβόνας και είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξει πρόοδος εδώ για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό. Ήδη είχαμε δεκάδες τέτοιες πρωτοβουλίες στο εξωτερικό και με την ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας ε, θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις παγκόσμιες ευθύνες μας καλύτερα, πράγμα άλλωστε που αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται καλύτερο συντονισμός για τις καινούργιες απειλές, ε, ε κυβερνοέγκλημα, ε, εμπορία ανθρώπων. Ε, χρειάζεται να υπάρξει οικονομία κλίμακος και αποφυγή των επικαλύψεων. αρκετοί αγορητές ε, μίλησαν και για τον μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο της βιομηχανίας άμυνας στην ευρωπαϊκή οικονομία και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Μεγάλες επενδύσεις και προσπάθεια πρέπει να γίνουν για την καλύτερη συνεργασία και συντονισμό σε αυτό το τομέα. Ε, όταν έλαβα το λόγο προηγουμένως είπα ότι πρέπει να συνεργαστούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ΝΑΤΟ, τον ΟΣΑ και άλλους τον ΟΑΣΕ και άλλους. Ε, πολλοί ομιλητές ε, ανέφεραν ε, τα προβλήματα επικαλύψεων με τα αεροσκάφη, τις φρεγάτες σκάφη και σε άλλους τομείς εξοπλισμού. Γιατί έχουμε κατακαιρματισμένες αγορές και δημόσιες συμβάσεις. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα εξετάσουμε να τα λύσουμε για να ωφεληθούμε από οικονομίες κλίμακος και να συνενώσουμε δυνάμεις και πόρους ούτως ώστε να έχουμε καλύτερα προϊόντα, να συνενώσουμε τους ε, ε, περιορισμένους μας πόρους. Νομίζω ότι το θέμα αυτό πρέπει να προσεχθεί πολύ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι στην ημερήσια διάταξη και πρέπει να επιτύχουμε απτή πρόοδο. Ε, συμβατικές ρυθμίσεις. Εδώ πρέπει να συνεχίσω με τη συζήτηση γιατί η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ε, συμβατικές ρυθμίσεις δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητή και νομίζω ότι θα πρέπει μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσουμε περισσότερες εξηγήσεις στο μέλλον γιατί όλοι συμφωνούμε και το είδα μέσα από την μεγάλη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο six και ΤΟΥΠΑΚ ότι αυτό που χρειάζεται είναι να βελτιώσουμε την οικονομική διακυβέρνηση. Είδαμε ε, πώς εξελίσσονταν τα ευρωπαϊκά εξάμεινα και πώς βελτιώνονται κάθε χρόνο. Τώρα, για τις ε, συμβατικές ρυθμίσεις νομίζω ότι θα πρέπει να προσθέσουμε το στοιχείο της οικονομικής υποστήριξης, της κινητοποίησης για μέτρα που καμιά φορά είναι δαπανηρά και δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν. Βεβαίως θέλουμε να σεβαστούμε απόλυτα το δικαίωμα δημοκρατικού ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, γιατί οι προτάσεις για αυτές τις συμβατικές ρυθμίσεις πρέπει να προέλθουν από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Θα προτείνουν εκείνα τι θέλουν να κάνουν. Ε, να αναλάβουν δέσμευση υπέρ των μεταρρυθμίσεων και πρέπει να δούμε τρόπους για να χρηματοδοτήσουμε τις μεταρρυθμίσεις αυτές στο μέλλον. Βέβαια, οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να σέβονται απόλυτα όλα τα καινούργια στοιχεία που προσθέσαμε στην κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Και η σύγκληση είναι ένας παράγον κλειδί στην οικονομική διακυβέρνηση και την ε, εφαρμογή, υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Εξαμήνων. Τέλος για την Τραπεζική Ένωση. Νομίζω ότι εδώ είμαστε σε κρίσιμη καμπή. Ε, υπάρχουν δύο τριμερείς διάλογοι σήμερα για την εγγύηση των καταθέσεων και την εξυγίανση και ανάκαμψη των τραπεζών, τη σχετική οδηγία και ελπίζομαι να υπάρξει πρόοδος γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να ολοκληρωθούν ε, αυτές οι δύο πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις πριν από τη ε, διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου. Πρέπει ε, να αρχίσει η νέα θητεία του Κοινοβουλίου με έτοιμη την Τραπεζική Ένωση. Κάποιοι αναφέρθηκαν στη συζήτηση για τον νέο μηχανισμό εξυγίανσης. Είναι δύσκολο αυτό. Το 114 λέει Κομισιόν είναι σωστή νομική βάση για όλα τα θέματα και το Ταμείο. Οι διαπραγματεύσεις όμως είναι πολύ δύσκολες και όπως ξέρετε οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών στο ΕΚΟΦΗΝ θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα και θα γίνει σκληρή δουλειά για την τελική συμβιβαστική λύση και τον σημαντικό ρόλο που έχει να παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία αυτή. Παράλληλα όμως πιστεύω ότι πρέπει να ομολογήσουμε ότι αυτή είναι μια διαδικασία σύσταση, συγκρότηση ενό συστήματο και αυτό παίρνει χρόνο. Ξεπεράσαμε σημαντικά εμπόδια. Πρέπει τώρα να, ε, αρχίσει, να ξεκινήσουμε το μηχανισμό, γιατί αυτό θα είναι σημαντικό μήνυμα στι χρηματοαγορέ, σημαντικό για τι επιχειρήσει, του πολίτε, που θα δείξει ότι επιτέλου κλείσαμε όλε τι τρύπε, όλα τα κενά και επιτέλους το τραπεζικό σύστημα ε, υπόκειται στο σωστό έλεγχο, ε, εδράζεται επί στέρεων θεμελίων και αυτό θα μας επιτρέψει να ξαναρχίσουμε τη χρηματοδότηση της οικονομίας που είναι ένα από τα βασικά προβλήματα γιατί η μεγέθυνση δεν ε, επιταχύνεται πράγμα που τόσο πολύ θα θέλαμε όλοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Πρόεδρε. Ευχαριστώ Μάρος. Θα ολοκληρώσουμε την συζήτηση με την παρέμβαση του Υπουργού Λεσκεβίτσιου, ο οποίο θα μας μιλήσει εξ του Συμβουλίου και της Προεδρίας του. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, είμαι ευγνώμων σε αυτούς όπου συμμετείχαν στη συζήτηση. Άκουσα ε, με πάρα πολλές απόψεις και ε, θα ληφθούν υπόψη στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, του οποίου προεδρεύουμε. Πολλοί από εσά ανέφεραν την Ουκρανία και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Ως ε, υπουργό ε, πάρα πολύ ε, νωρίς το πρωί και χτες το βράδυ είδα τους διαδηλωτές και πώς ακολούθησε ένα μη ευρωπαϊκό δρόμο το θέμα αυτό βλέπουμε τη δράση αυτή ότι δεν σέβεται την ελευθερία, την ελευθερία του συναθρίζεσθε, την ελευθερία του λόγου που βρίσκονται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αξιών. Ε, είμαστε ευγνώμονες στην ύπατη εκπρόσωπο διότι προσπαθεί να βρει μια πολιτική λύση για το θέμα αυτό στο Κίεβο με άμεση εμπλοκή προσωπική. Ο πρόεδρος Μπαρόζο είπε ότι σε αυτές τις δύσκολες ώρες δεν μπορούμε να αφήσουμε το λαό αυτό μόνο του και θα ήθελα να ευχαριστήσω το γεγονός ότι μία, ένα ψήφισμα θα ψηφιστεί αύριο σε σχέση με το θέμα αυτό. Τέλος, σχετικά με την Ουκρανία, όπως έλεγα κατά τη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης, είναι εξίσου σημαντικό να είμαστε παρόντες. Απλώς να είμαστε παρόντες, να επιδείξουμε ότι ο λαός αυτός δεν έχει μείνει μόνος. Μερικοί βουλευτές ο κύριος Βόμποντα και η κυρία Πέρες ανέφεραν ιδιαίτερα την κοινωνική διάσταση. Βεβαίως είναι σαφές ότι η ανάπτυξη μόνη της δεν πρόκειται να διορθώσει την κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η ανάπτυξη θα πρέπει να δημιουργεί θέσεις εργασίας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της κρίσης και να αυξήσουμε ε, τις ε, προσπάθειες για να υπάρχει εξισορρόπηση ανάμεσα στις οικονομικές και στις κοινωνικές διαστάσεις καλή ε, λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης χρειάζεται ούτω ώστε με ισορροπημένο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της ανεργίας και της κοινωνικής ανισορροπίας. Μια ε, δυνατή ε, κοινωνική διάσταση θα δώσει τις καλές προτεραιότητες στην πλήρη απασχόληση. Η κοινωνική διάσταση θα πρέπει να οικοδομηθεί γύρω από μια προσπάθεια ούτω ώστε να υπάρχει απασχόληση, ε, εκπαίδευση και κατάσταση χωρίς αποκλεισμούς. Τα περισσότερα κράτη-μέλη είναι υπέρ της εισαγωγής ε, να έχουμε μια βαθμολόγηση σχετικά με τα θέματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ένα μέσο αυτό, το μέσο αυτό του πίνακα βαθμολόγησης θα μας επιτρέψει να δούμε τι γίνεται με την κοινωνική πολιτική και την απασχόληση. Επίσης, τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν την πρόταση βελτίωσης των μηχανισμών, ούτω ώστε να υπάρχει ε, συντονισμός με τα εθνικά επίπεδα, ανάμεσα στο ευρωπαϊκό και στα εθνικά επίπεδα. Κύριε Επίτροπε, ο κύριος Επίτροπος ανέφερε το θέμα των αποταμιεύσεων, την οδηγία. Χθες δεν είχαμε ακόμα πολιτική συμφωνία. Θα ήθελα ότι η Προεδρία δεν εφίστη καμιά προσπάθεια για να έχουμε μια τέτοια οδηγία πριν από το τέλος του έτους όπως ζητά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν ε, στην ατζέντα της, ε, του ΕΚΟΦΗΝ το Δεκέμβριο, αλλά δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία στο στάδιο αυτό λόγω ορισμένων επιφυλάξεων ορισμένων κρατών μελών. Η έκθεση η οποία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παρουσιάσει το αποτέλεσμα των συζητήσεων του ΕΚΟΦΗΝ και τότε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει τι σήμα, τι μήνυμα θέλει να στείλει σχετικά με την συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί σε αυτό το φάκελο. Ο κύριος Βαν Άρντεν και η κυρία Γκόμες ανέφεραν ορισμένα συγκεκριμένα ε, σημεία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Θα ήθελα να πω το εξής. Αυτή την εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, θα μπορέσει να ψηφίσει αποτελέσματα για να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα στον τομέα αυτών σχετικά με την πολιτική της άμυνας στον κυβερνοχώρο ε, και τη στρατηγική θαλάσσιας ασφάλειας και να αυξήσουμε τις αδυνατότητες ε, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη συστημάτων αεροπορικών ε, μέσα στα πλαίσια μέχρι το 2025 και επίσης ανάπτυξη για ε, την δυνατότητα αερομεταφοράς για την δορυφορική επικοινωνία, ανάπτυξη ενός χάρτη πορείας όπως και σχεδίων για να βελτιώσουμε την στρατιωτική και μη στρατιωτική συνεργασία ε, για την στρατηγική στον κυβερνοχώρο. Μερικοί από εσά ανέφεραν τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ επίσης, Ευρωπαϊκή Ένωσης ΝΑΤΟ. Θα ήθελα να τονίσω ότι το ΝΑΤΟ είναι βασικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να το τονίσει αυτό στα πορίσματα σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Το Συμβούλιο θα ήθελε να υφετηθούν και άλλα πρακτικά ε, μέτρα για συνεργασία με το ΝΑΤΟ με συνολικό στόχο να έχουμε μια πραγματική σχέση με την οργάνωση αυτή που θα περιλαμβάνει επίσης το να αποφεύγουμε την, ε, το τις επικαλύψεις. Η επόμενη εβδομάδα η συνάντηση θα καλύψει διάφορα θέματα, ένα ολόκληρο φάσμα ε, θεμάτων που άπτονται των ε, συμφερόντων των πολιτικών των πολιτών. Ε, θα πρέπει να βοηθήσουμε ε, τη οικογένειες ε, ούτως ώστε να έχουν ένα περιβάλλον ασφαλέστερο. Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι ένας διαφορετικός τρόπος εξασφάλισης από την αβεβαιότητα την οικονομική και τον φόβο της μακροχρόνιας ανεργίας. Η Τραπεζική Ένωση ε, σκοπεύει να προστατεύσει την ζωή από μια, ε, των πολιτών από μια άλλη ε, οικονομική κρίση, ούτως ώστε να έχουμε ευρωστία των ε, τραπεζών στις οποίες εμπιστευόμαστε τις οικονομίες μας. Επίσης το θέμα της μετανάστευσης από την Μεσόγειο αποβλέπει στο να προστατεύσει όσους κινδυνεύουν και αναζητούν καλύτερη ζωή τους οφείλουμε ε, να αποφευχθεί ε, η επανάληψη της καταστροφής ε, που είχαμε τον Οκτώβριο. Θα έχουμε τις ευρωεκλογές του χρόνου και θα μπορούμε να επισημάνουμε τα θέματα αυτά όπου η Ευρώπη κάνει την διαφορά σε συνεργασία και με αλληλεγγύη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Έχουμε δεχτεί τέσσερα ψηφίσματα, τέσσερα προτάσεις, ε, τέσσερις προτάσεις ψηφισμάτων για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Ε, ένα από το ΕΛΚ, ένα από τους σοσιαλιστές, ένα από τους φιλελεύθερους και ένα από την ΚΟΕ, την Ευρωπαϊκή Νοτική Αριστερά. άλλο ένα πίσω από τους πράσινους και ένα από τους